Guten Morgen, guten Morgen, good morning. Good morning, liebe Kolleginnen und Kollegen. Καλημέρα, συνάδελφοι. Einer ganzen Reihe von... Έχουμε μια ολόκληρη σειρά ψηφοφοριών, αλλά θα ξεκινήσουμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αν συμφωνείτε, θα ήθελα καταρχήν να σας πω ότι εν ώψη της κατάστασης στην Ιαπωνία και επειδή είμαστε υπεύθυνοι για θέματα περιβάλλοντος, για θέματα δημόσιας υγείας, για θέματα τροφίμων και βεβαίως δημόσιας υγείας θέλω να εκφράσω την λύπη μας για αυτά που συνέβησαν και μετά τον σεισμό, το τσουνάμι και κυρίως την ε, κατάσταση η οποία ακόμα δεν είναι σαφής όσον αφορά τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στην ε, Φουκοσίμα. Διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά ότι η φύση είναι πιο δυνατή από τον άνθρωπο. Αυτό είναι κάτι που πολλές φορές το έχουμε πει εδώ στην Επιτροπή μας όταν κοιτάμε τις αλλαγές του κλίματος, όταν βλέπουμε τα φυσικά φαινόμενα και άλλες έντονες αντιδράσεις της ε, φύσης που πλήττουν τον άνθρωπο, διαπιστώνουμε ότι δεν ελέγχουμε τα πάντα. Και νομίζω ότι σήμερα μπορούμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας προς τους πολίτες ε, της ε, Ιαπωνίας και να πούμε ότι η διαχείριση αυτής της καταστροφής έγινε με εξαιρετικό τρόπο από την Ιαπωνία. Έχουμε στείλει εξάλλου δυνάμεις από την Ευρώπη για να βοηθήσουν να ξεπεραστεί αυτή η τεράστια φυσική καταστροφή. Γι' αυτό λοιπόν και θα προτείνω και μια αλλαγή της ημερήσιας διάταξης σήμερα το μεσημέρι. Ο Γκίντερ Έντιγκερ θα έρθει γιατί θέλουμε να μας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ευρώπη όσον αφορά τις ε, 143 ε, πυρηνικές μονάδες που έχουμε στη χώρα μας, στην Ήπειρό μας, ε, συγγνώμη. Σας ε, παρακαλώ να είστε ακριβείς, γιατί η Πατρίσια Εσπινόζα θα είναι εδώ με το πολύ σημαντικό θέμα Κανκούν και την επόμενη συνδιάσκεψη για το κλίμα με πρέσβεια του Μεξικού. Επίσης υπάρχουν κάποια σημεία που πρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε το 15 και το 16. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για ερωτήσεις, παραδείγματο χάρη, ενδεχομένως ερωτήσεις ενός λεπτού, αλλά πρέπει πραγματικά να είμαστε ακριβείς και σύντομοι. Μετά τον κύριο Έτιγκερ, να πάμε στο σημείο 23. Ε, αν συμφωνείτε, καθότι η κυρία Ζόμερ, η συγγήτρια, θα ήθελε να μας κάνει την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα. Κατόπιν μπορούμε κάποια σημεία να τα αναβάλουμε για τις 11-12 ε, Απριλίου την επόμενη ε, έχουμε το θέμα της εντολής για τον τριμερή διάλογο. Όχι. Έχουμε επίσης τον αριθμό κλήσης 112. Αυτό να αναβληθεί επίσης. Αύριο τώρα. Το σημείο 25. ΑΕΠ και πέρα από αυτό, Beyond GDP, αυτό να μετακινηθεί μετά το 26 μετά δηλαδή τη διαχείριση καυσίμων διαρρεδιών αποβλήτων. Αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρουμε όλοι ότι τις τελευταίες μέρες η κατάσταση άλλαξε πολύ στην ενεργειακή αγορά. Και ξέρουμε ότι θα πρέπει να κάνουμε μια επαλήθευση των ενεργειακών μας πόρων, κυρίως ό,τι αφορά τα πυρηνικά. Καλό θα ήταν λοιπόν για ακόμα μία φορά να αναρωτηθούμε αν θα πρέπει να έχουμε δύο benchmark. Ένα για το φυσικό αέριο και ένα άλλο για τον άνθρακα. Όχι με βάση όμως τα παλιά συστήματα και τις παλιές τεχνολογίες, με βάση τις νέες τεχνολογίες, ούτως ώστε να μην ξαναβρεθούμε σε μια κατάσταση όπου μας λείπει η ενέργεια. Μπορούμε ακόμα να κάνουμε παληθεύσεις και να έχουμε δύο τέτοια μέτρα συγκριτικής, μέτρα συγκριτικής αξιολόγησης. Σας παρακαλώ λοιπόν ε, υποστηρίξτε αυτά τα δύο σημεία που είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας και για το σύνολο της Ευρώπης. Εδώ αναφέρεστε στο σημείο 5. Ναι, είσαστε ήδη στο 5 ψηφοφορία για το benchmarking. Bitte? για το σημείο 2 της ψηφοφορίας. Το σημείο 2 της ναι, ναι, ψηφοφορίας. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Σας άκουσα. Σας άκουσα. Δεν υπάρχει δυνατότητα εδώ να σας απαντήσω. Μπορούμε απλώς να πούμε ναι ή όχι στο ψήφισμα. Συνεχίζουμε λοιπόν, λέει ο Πρόεδρος, με δύο ανακοινώσεις. Άννα Ρόσπα, η οποία άλλαξε πολιτική ομάδα έγινε μέλος της ομάδας η αυτή. Και τώρα τη βλέπω να κάθεται ειρηνικά και ήσυχα δίπλα στους συναδέλφους από την ομάδα της. Έχουμε και ένα νέο συντονιστή για την ομάδα αυτή, Ρώση. Και θα είναι και παρόν στην συνάντηση των συντονιστών. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι υπάρχουν κάποια εργαστήρια όσον αφορά τις ε, εκπομπές 22 Μαρτίου το πρωί. Είστε όλοι καλεσμένοι. Επίσης μας έχει καλέσει η Επιτροπή Ήτρε, Βιομηχανίες για τις ανανεώσιμες τεχνολογίες την ίδια μέρα, 22 Μαρτίου το απόγευμα. Αυτά όσον αφορά τα εργαστήρια και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Συμφωνία προστασίας και αηφόρου ανάπτυξης της περιοχής του Πάρκου Πρεσπών. Ο κύριος Αρσένης είναι εισηγητής και θα του δώσω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είχαμε χρόνο να το συζητήσουμε αυτό στην Επιτροπή, γιατί θέλαμε να προχωρήσουμε με την ψηφοφορία. Έτσι λοιπόν, έχει, έτσι ώστε να εγκριθεί καιρό και να τεθεί σε ισχύ το περιβάλλον, δεν έχει σύνορα. Εδώ μιλάμε για ένα υγροβιότοπο που ανήκει σε τρία κράτη, την ε, Ελλάδα, τη Φιρόμ και την Αλβανία υπήρξε μια συμφωνία για τη μέτρα κοινή προστασία σε αυτό το σημαντικό που είναι και περιοχή Natura 2000 αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται και από τη Σύμβαση Ράμσα. Έτσι λοιπόν η συζήτησή μας εδώ και η ψηφοφορία μας επιτρέπει την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αρσένη. Ψηφίζουμε υπέρ. κατά αποχές ομόφωνα. όπως μου λέει η γραμματεία, πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αν λοιπόν έχετε όλοι τις κάρτες σας, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, γιατί έτσι γίνεται συνήθως αυτού του είδους ψηφοφορία. Αρχή της ψηφοφορίας. μία επιπλέον ψήφος. Τέλος. 57 υπέρ, κανείς κατά. Ομόφωνα λοιπόν εγκρίθηκε, συγχαρητήρια. Και περνάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 8 παραγραφός 2. Καθορισμός μεταβατικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εναρμόνιση δωρεάν κατανομής αδειών εκπομπής αερίων δείκτες αναφοράς, benchmarking. Η πρόταση ψηφίσματος έχει υποβληθεί, μάλιστα δύο είναι, Φιλίπ Ζεβά, Αγιούζο και άλλοι, Ήπνερ. Ψηφίζουμε λοιπόν, αρχή της ψηφοφορίας για το πρώτο κείμενο. Πάλι μία ψήφος παραπάνω βγαίνει. Jetzt ist gut. Τέλος της ψηφοφορίας. 13 υπέρ, 60 κατά, 4 Αποχές απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στο δεύτερο ψήφισμα. Τσιμένσκι. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Εννέα υπέρ. 44 κατά, δύο εποχές Απορρίπτεται και αυτό. Και τώρα προχωρούμε. Ήθελα να πω ότι ο κύριος Κυλακάκης, όσον αφορά το benchmarking, έχει αναφερθεί στην παραγωγή δέσει στα ελληνικά νησιά και περνάμε στο σημείο 6. Όπως ε, βλέπετε, πρόκειται για το θέμα DHA στο γάλα για βρέφη. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος της ψηφοφορίας. Δεκατρεις... Συγγνώμη, 30 υπέρ. 28 κατά. Εγκρίνεται. Σημείο 7. Απαλλαγή. Γενικός προϋπολογισμός. Απαλλαγή 2009. Γενικός προϋπολογισμός, τμήμα 3, Επιτροπή. Επαναλαμβάνω σημείο 7 της ημερησίας διάταξης. Πολλές τροπολογίες. 1. Τόλμας Ούλμα. Υπέρ. Τροπολογία 1. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2. Λάμστορφ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τρία Με προφορική τροπολογία και ξεχωριστή. Πρώτο τμήμα με την προφορική τροπολογία ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Και τώρα ψηφίζουμε για την τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά, αρχή της ψηφοφορίας. Πάλι ένας επιπλέον στους σοσιαλιστές. Ψηφίσαν όλοι. Τέλος. 49 υπέρ. 5 κατά. Μία αποχή. Συγχαρητήρια. Γιούτα Χάουκ. Μακάρι όλες οι ψηφοφορίες να έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σημείο 8. Πρόκειται για την απαλλαγή 2009 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος. Τροπολογία 1 Είχε αποσυρθεί. 2. Αλέξανδρ Λάμστορφ. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τρία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, αρχίζουμε. Τέλος. 51 υπέρ, κανένας κατά, 6 αποχές. Μεγάλη εμπιστοσύνη για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Η επόμενη ψηφοφορία, Ευρωπαϊκός Οργανισμός φαρμάκων. Τροπολογία 1, Τόμα Ούλμαν. Υπέρ. Κατά. απόχέ. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. απόχέ. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 4 καταπίπτει. Ψηφίζουμε και την τροπολογία 4, το πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4, δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5, υπέρ. Κατά Αποχές. Εγκρίνεται. 6. Αποσύρθηκε. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίψτε. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζουμε. τελείωσε η ψηφοφορία. Και τώρα ψηφίζουμε για το επόμενο θέμα, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Τροφίμων, ΕΦΣΑ. Ψηφίζουμε την τροπολογία 2, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Καταπίπτει η 1 και πάμε στην τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 4 έχει αποσυρθεί. 5 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για την ΕΦΣΑ, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Τέλος. 45 υπέρ, 6 κατά, 6 εποχέ. Συγχαρητήρια. Και τώρα περνάμε στον Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, ξεχωριστή ψηφοφορία στην παράγραφο 2. Το πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Ξεχωριστή ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία να έχει αποσυρθεί. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 2. Τέλος. Απορρίπτεται. 27 υπέρ, 29 κατά. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 5 υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. 43 υπέρ 4 κατά 7 αποχές. Συγχαρητήρια. Και τώρα περνάμε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, η τρία έχει αποσυρθεί, η 4 υπέρ, κατά, η πέντε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος της ψηφοφορίας. 49 υπέρ. Κανείς κατά 7 αποχές. Γιούτα Χάουγκ. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά για την εξαιρετική εργασία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα είμαστε στο σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης. πράσινη βίβλος της Επιτροπής Προστασία Δασών και σχετική πληροφόρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προετοιμασία των δασών εν ώψη της αλλαγής του κλίματος. Έχω μια καταπληκτική λίστα εδώ για την ψηφοφορία. Ο κύριος Αρσένης έχει το λόγο. Thank you very much, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συζητητές ε, και τη γραμματεία και ε, όλους τους συμβουλούς από όλα τα κόμματα στην ε, πολύ καλή δουλειά που έγινε στο να καταλήξουμε σε 48 συμβιβασμούς, ορισμένες ε, τροπολογίες, αλλά έχουμε ένα σημαντικό αριθμό συνένεσης μεταξύ των κομμάτων επί των συμπερασμάτων και του συμβιβασμού στα οποία καταλήξαμε. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους για την πολύ καλή δουλειά. vielen Dank. Ευχαριστούμε πολύ. Όντως μια μεγάλη, ένας μεγάλος αριθμός συμβιβαστικών τροπολογιών. Ψηφίζουμε. Συμβιβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά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 Αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. 30. Συμβιβαστική 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έχουμε πολλές ακόμα. Όλες πρέπει να τις ψηφίσουμε ξεχωριστά. Υπάρχουν ορισμένες ε, ενωπημένες μεταξύ αυτών. Ε, δεν με πειράζει αν ε, τις ψηφίσουμε και όλες μαζί. Αλλά η κάθε μία περιλαμβάνει σχεδόν 10 τροπολογίες στο συμβιβασμό. Πρέπει όλοι οι συνάδελφοι να γνωρίζουν ότι είχαμε 370 τροπολογίες για την έκθεση αυτή. Έτσι λοιπόν τώρα κερδίζουμε πάρα πολύ χρόνο. 30 φορές αποδείχθηκε ότι είναι καλός ο συμβασμός. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και στις υπόλοιπες σε μπλοκ. Στις 17-18 υπόλοιπες. 31, συμβεβαστική 31 με 48, υπέρ, κατά, αποχές, με τρομερή πλειοψηφία εγκρίθηκαν. Λοιπόν, τι μας μένει να ψηφίσουμε. 99, τροπολογία 99, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 100, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 101. 101 υπέρ. Να ελέγξουμε την 100. Ωραία. Ελέγχουμε την 100. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος. Είναι σαφές το αποτέλεσμα. Εγκρίνεται. 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 102. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.

Όλες αυτές είναι ίδιες. Υπέρ. Κατά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος. Απορρίπτεται. Ναι. 125 υπέρ κατά αποχές δεν σηκώνουν τα χέρια φιλελεύθεροι δεν καταλαβαίνω τι κάνετε είστε υπέρ, είστε κατά 125 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται, αλλά ελέγχουμε παρόλα αυτά. Τέλος. Απορρίπτεται. Άξιζε. 123. Υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. Α, ελέγχουμε. Τέλος, απορρίπτεται. 127 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 126 είναι γλωσσική, 130 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 131 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 138 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στη σελίδα 11, 158, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 159 τώρα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 166 έχει αποσυρθεί. 172. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 173 Έλενα ο άναν τον Έσκο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ήτρε 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 174 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 186 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Σελίδα 15 ήτρε 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 200. Πέντε, Κλάς και Σνέλχαρτ. Υπέρ. Μάλλον. Υπάρχει και μία προστίκη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. Κοιτάξτε το αποτέλεσμα. Αποσύρεται η 207. 206 με μία προσθήκη υπέρ. 206 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 211 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 212 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την 212. Ψηφίζουμε. Τέλους ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έξι άτομα όμως δεν ψηφίζουν ηλεκτρονικά. Σημαίνει ότι δεν έχετε κάρτες. 2.13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 έχει αποσυρθεί, 2.22, 2.23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 227 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 229 υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη 229. Τέλος. Εγκρίνεται. Η 230 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 235 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 241 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 248 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 251 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 252 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 17 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 254 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 255. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 257. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 258 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 261 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ήτρε 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ήτρε 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 262 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 263 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 266 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. 266 αρχή της ψηφοφορίας τέλος Εγκρίνεται η 266. Και μετά είμαστε στη σελίδα 25 ή 310 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 259 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. άγρι 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 294 με προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 296 με προφορική υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και Ελέγχουμε την 296. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Και τώρα πάμε. Η, η τροπολογία 13 έχει αποσυρθεί. Πάμε στη 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 έχει αποσυρθεί. 19 ή 34 36, το πρώτο τμήμα της 36. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα της 36, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 38, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 39, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σχεδόν λοιπόν, τελειώσαμε. 66. 66 στη σελίδα 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ όχι όχι 75 συγγνώμη υπέρ 75 Θεόδωρος Κυλακάκης υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Είναι ήδη 78, 79, 80, 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α, να το ελέγξουμε αυτό το τελευταίο αποτέλεσμα. 78 έως 82. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος. Απορρίπτεται. Δεν έφτασε. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά Εποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά Εποχές εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 89 και 90 μαζί, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκαν. 93 Α, όχι, πρώτα ελέγχουμε το 89-90. 89-90 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος, εγκρίνονται. Οι 93 και 92 καταπίπτουν και ψηφίζουμε την 94 υπέρα κατά, αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Και φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. 53 υπέρ 6 κατά καμία αποχή συγχαρητήρια στον ε, Κρήτον Αρσένη και σε όλους όσους στήριξαν αυτήν την ε, προσπάθεια. Ελπίζω να φτάσουμε σε μια πράσινη βίβλο για την προστασία των δασών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πραγματικά Πρόκειται για το 1 τρίτο της επιφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά αυτή την πράσινη βίβλο. Ωραία. Έχουμε φτάσει και στο σημείο 14. Τροποποίηση της οδηγίας του 2025 όσον αφορά τις διατάξεις για τους κινητήρες που διατίθενται στην αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου συστήματος. Εμένα εδώ λέει κινητήρες, αλλά φαίνεται ότι πρόκειται για τρακτέρ. Στα γερμανικά, λέει ο πρόεδρος, διαβάζω κινητήρες. Ίσως πρόκειται για λάθος. Ξεκινάμε λοιπόν με την επεξεργασία του θέματος αυτού και είμαστε στην τροπολογία 20 και 21. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές δεν πέρασε. Απορρίπτηκαν αυτέ οι δύο τυπολογίες. 22. 4 έχουν αποσυρθεί. 34 του Σαλβατόρε Ταρταρέλα, του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 3, Consolidated Amendment, τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Και συνεχίζουμε με την τροπολογία 38 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Η 9 έχει αποσυρθεί, η 39 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 7 έχει αποσυρθεί. Η 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 8 έχει αποσυρθεί. Η 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 9 έχει αποσυρθεί. Η 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 10 έχει αποσυρθεί. Πάμε στη 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 11 έχει αποσυρθεί. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 12 έχει αποσυρθεί. Και πάμε στο παράρτημα 1, τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 έχει αποσυρθεί. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 έχει αποσυρθεί. 52 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16 έχει αποσυρθεί. Τραν 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 17 έχει αποσυρθεί. 18 επίσης. 54 ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Η 19 έχει αποσυρθεί και τώρα πάμε στην τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Πίτερ Λίζε 25 ψηφίζουμε την 25 ποιος είναι υπέρ κατά ηλεκτρονική ψηφοφορία 25 Τέλος. Εγκρίνεται 25. Ένα έχει αποσυρθεί. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Τραν 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. απορρίπτεται 2. Τραν 2. Και κατόπιν πάμε στην τροπολογία 1, consolidated κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε στην τροπολογία 29. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Δεν μπορώ να δω. 29 του Πίτερ Λίζε. Ποιος είναι υπέρ. Τώρα σας βλέπω. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 33 έχει αποσύρθει και πάμε στην τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Τέλος. Και εδώ ψηφίζαμε για το σχέδιο. Πέντε αποχές. Γρίθηκε και τώρα πάμε στο σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Παρόλα αυτά, ναι, ψηφίζουμε αρχή της ψηφοφορίας, καφές, τσάι, όλα μαζί. Λείπουν, λείπουν, λείπουν. Δεν ψήφισαν όλοι. Κάντε μια προσπάθεια. Α, τώρα πάνε όλα καλά. Τέλος της ψηφοφορίας. 45 υπέρ, 5 κατά, 6 αποχές. Συγχαρητήρια, Σαλβατόρε Ταρταρέλα. Ήταν δύσκολο και περίπλοκο το θέμα αυτό και καταφέραμε να το στηρίξουμε. Προχωράμε στο επόμενο σημείο. Από τα τρακτέρα πάμε στους κινητήρες. Το επόμενο σημείο της ημέρης και διάταξης είναι το 15. Ήταν η Σύρπα Πίτι Κάινεν εισηγήτρια και ψηφίζουμε. Τροπολογίες 17, 18 για την ε, αναπομπή στην Επιτροπή. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκαν. Η 19 έχει αποσυρθεί έτσι κι Και πάμε στα άρθρα. Τροπολογία 8 έχει αποσυρθεί. Η 50 και 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 52 και 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 54. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτονται. 55 και 56. Α, για έλεγχο. Καλά, ε, εντάξει, δεν είναι ίσως δικαιολογημένο, αλλά το δέχομαι. Ελέγχουμε την 54. Τέλος. Εγκρίνεται. Είχα πει ότι απορρίπτεται. Ναι. Ναι. 55, 56. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 57 και 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 60. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα πάμε στην τροπολογία 11. Ποιος είναι υπέρ της 11. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66 και 68 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. 66 και 68. Ελέγχουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. Ε, πάμε στην τροπολογία 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 72 και η 73. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Και 74. Εξάλλου έπρεπε να είχαμε ψηφίσει μαζί. 75 ε, και 11. Υπέρ. Α, όχι, αυτό καταπίπτει. Και η 76. Α, τραν 4. Ψηφίζουμε την τραν 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 80 και 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 88 ποιος είναι υπέρ κατά α συγγνώμη συγγνώμη ξέχασα την 10 πριν την 88 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε την 88 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 5, τροπολογία 5 ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 4, τροπολογία 4 ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 4 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 98. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 15, η 99, η 100 και η 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στη σελίδα 8, 111 και 112. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκαν. Και τώρα πάμε στη τραν 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 113 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία 20. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε την 25. Τέλος. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία 3. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 5 καταπίπτει. Και μετά έχουμε την 38 και την 39. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Η 6 έχει αποσυρθεί. Η 41 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 6. 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε η 6. Και τώρα φτάσαμε στην τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το σχέδιο έκθεσης αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. 48 υπέρ 7 κατά 2 αποχές. Και τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Τέλος. 51 υπέρ, 5 κατά, 2 αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια, στους κοιόδης και σε όλους όσους βοήθησαν σε αυτήν την δύσκολη προσπάθεια συμβιβασμού. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Σύρπα, έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Ε, κοιτάξτε, εδώ κάναμε ουσιαστικά μια πρόβα τακτικής. Θέλω να δράξω την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους στην ομάδα μου και τους σκιώδεις εισηγητές και τους λοιπούς συναδέλφους που συνέσφεραν σε αυτά τα καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ε. Και εμείς ευχαριστούμε. Όντως είναι πολύ σημαντικό να ακούμε προσεκτικά και να ακολουθούμε την γραμμή που μας προτείνεται. Το επόμενο σημείο είναι το 16. Ένωση καινοτομία. Μεταμορφώνοντας την Ευρώπη για ένα κόσμο μετά την κρίση. Ο Ζωάου Φερέρα είναι ο εισηγητής. Ψηφίζουμε. Τροπολογία 1. Αρσένης. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2. Έχει αποσυρθεί. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3. Όχι. Συγγνώμη. Ψηφίσαμε τη 3. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απο... Ε, εγκρίνεται. Συγγνώμη. 5. Υπέρ. Κατά αποχές. Το ΕΛΚ κάνει, δεν είδα. Στην 5. 5. Υπέρ. Ξαναψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 5. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7. Υπέρ συγγνώμη, 9 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12. Καταπίπτει 12. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. η 11. 14. Α, να ελέγξουμε την 11. Η έντιτε στρέλα ζητάει έλεγχο για την 11. Έχουμε ξεκινήσει. Τέλος. Απορρίπτεται η 11. Και ψηφίζουμε τη 14. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 16 έχει αποσυρθεί ψηφίζουμε την 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 18 Ξεχωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα πρώτα. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 20 υπέρ. Α, να ελέγξουμε το 19. Ψηφίζουμε λοιπόν το 19. Τέλος. Εγκρίθηκε. Το 19 εγκρίθηκε. Και περνάμε στην τροπολογία 20. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 21. Το πρώτο τμήμα πρώτα. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 22 έχει αποσυρθεί 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το 25 το πρώτο τμήμα πρώτα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 26. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 27. Υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 28. Το πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Πρώτο τμήμα 28. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα του 28. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τέταρτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 29 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 30 ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 31 το πρώτο τμήμα υπέρ, Ο εισηγητής. Πρόεδρε, εγώ ήθελα να αποσύρω το αίτημα της χωριστής ψηφοφορίας, επομένως να ψηφίσουμε το σημείο αυτό στο σύνολό του και ήθελα να προτείνω ψήφο κατά. Υπέρ. Κατά. αποχές, έλεγχος. Τέλος. Απορρίπτεται. 32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 47 υπέρ, κανείς κατά, 8 αποχές. Συγχαρητήρια Ζωάου Αφερέρα. Πρόκειται για την Ένωση Καινοτομίας. Η τελευταία ψηφοφορία για σήμερα το πρωί είναι το σημείο 17. Πρόγραμμα στήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής η συγγήτρια είναι η Κορίν Λεπάζ. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 και 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5. Το πρώτο τμήμα του 5. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα του 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 με μία προσθήκη του κυρίου Τρεμόπουλου υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 28. Το αποτέλεσμα είναι 30 κατά 26 υπέρ. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 30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 16. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτό εγκρίνεται. 40. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 42 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 18. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 43 με την προσθήκη που βλέπετε, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Δύο ίδιες τροπολογίες, 44-45, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 46 ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 47 έχει αποσυρθεί. Ψηφίζουμε τη 48, 49, 50, ποιος είναι υπέρ. 48, 49, 50, κατά. Αποχές απορρίπτονται. 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 20 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίθηκε και 20. Πάρα πολύ καλή γυμναστική κάναμε σήμερα το πρωί, σηκώνοντα και κατεβάζοντας τα χέρια. Ψηφίζουμε για τελευταία φορά, αρχή της ψηφοφορίας, τέλος 53 υπέρ, κανείς κατά και μόνο μία αποχή. Μεγάλη στήριξη, συγχαρητήρια στην εισηγήτρια κυρία Λεπάζ και σε όλους τους κοιόδους οι οποίοι βοήθησαν. Ευχαριστούμε επίσης και τη Γραμματεία για την εξαιρετική προετοιμασία αυτής της ψηφοφορίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο σας. Έχουμε κι άλλο ένα σημείο όμως. Ja, also wir sind bei dem Punkt 18. Είμαστε στο σημείο 18 Πρόκειται για μια προφορική ερώτηση για την Ολομέλεια. Ποιος είναι υπέρ αυτής της πρότασης για προφορική ερώτηση. Ποιος είναι κατά, ποιος απέχει, εγκρίνεται. Οπότε θα υποβάλουμε αυτή την ερώτηση στην Ολομέλεια για συζήτηση. Και περνάμε αμέσως στο σημείο 19. Yeah, Linda. Sorry, colleagues, we just adopted an oral question on task. Μόλις ε, υιοθετήσαμε την προφορική ερώτηση για τον ασβεστούχο, για τον ασφαλτούχο ε, άμμο θα γίνει μια ειδική ενημέρωση στο 5G1 στις 12.45. Ε, Υπάρχει και μια έκθεση επίσης μπροστά από το Κοινοβούλιο στην ε, πλατεία Λουξ, ε, στις 2 και 4 μπορείτε να ενημερωθείτε. Θα σας στείλω και θα τα βρείτε και, θα τα βρείτε και στα ηλεκτρονικά σας α, ταχυδρομεία όλα αυτά τα στοιχεία. Ναι, είναι κατά τη διάρκεια της μεσημερινής διακοπής μπροστά από το Κοινοβούλιο. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο όμως, Μπάς Έικουτ, πρόκειται για την ανάλυση επιλογών για την καταπέρα των 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκτίμηση του κινδύνου διαρροής άνθρακα. Έχουμε ένα έγγραφο εργασίας και σήμερα θα μιλήσουμε και θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης. Μπας Άικουτ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Μετά από τις ψηφοφορίες μπορούμε να χαλαρώσουμε και να ακούσουμε μια έκθεση. Για να δούμε τη συζήτηση που θα λάβει η χώρα είναι σαφές ότι στην έκθεση ζητά από την Κομισιόν να κάνει προτάσεις για να αυξήσει τις ε, κλιματικές φιλοδοξίες σε 3% μέχρι το 2020, το συντομότερο δυνατόν ε, και ή δυνατόν πριν το τέλος του 2011. Φυσικά μπορούμε να πούμε ότι μια μετακίνηση προς 40% θα ήταν πολύ πιο λογικό, αν λάβουμε υπόψη μας τα επιστημονικά στοιχεία, και αν υπάρξουν τροπολογίες προς αυτήν την κατεύθυνση θα τις υπερψηφίσω. Αλλά σε αυτή την έκθεση απλώς ζητάμε τη μείωση των ε, εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 30%. Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για να ζητούμε αυτή την αύξηση σε 30%. Καταρχάς, ε, υπάρχει μια κλιματική κρίση, θα έλεγα, με κατεπήγοντα χαρακτήρα. Οι επιστήμονες λένε ότι μέχρι το 2015 θα αυξηθούν οι εκπομπές και θα πρέπει η Ευρώπη να κάνει ό,τι μπορεί. Και το 20%, η μείωση κατά 20% δεν είναι αρκετή για να αντιμετωπίσουμε τις εκπομπές μέχρι το 2015 που θα αυξηθούν, θα φτάσουν στο ανώτατο όριο μέχρι το 2015. Ε, τα τελευταία τώρα χρόνια αυτά τα κλιματικά επιχειρήματα ε, έχουν γίνει πολύ σημαντικά. Και νομίζω ότι είναι και προς το συμφέρον μας να αυξήσουμε τις φιλοδοξίες. Αν δούμε τις εισαγωγές πετρελαίου, αυξήθηκαν κατά 70 ε, δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι. Και αν αυξηθούν η, εκπο... μείωση των εκπομπών από το 20% στο 30% μπορούμε να μειώσουμε το λογαριασμό μας μέχρι το 2020 για το πετρέλαιο κατά 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Αν ας πούμε ε, υποθέσουμε ότι η τιμή του βαρελιού θα είναι 88 δολάρια το βαρέλι. Φυσικά αν αυξηθεί το, η τιμή του βαρελιού θα έχουμε περισσότερα κέρδη. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο επιχείρημα για τις θέσεις απασχόλησης. Τον περασμένο μήνα ε, υπήρξε μία μελέτη που παρουσιάστηκε στην μόνιμη γερμανική αντιπροσωπεία που έλεγε ότι αν αυξήσουμε τις φιλοδοξίες μας για το κλίμα θα έχουμε επιπλέον 6 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Αυτό όταν ε, τον περασμένο Μάιο συνέταξε η Επιτροπή την ε, ανακοίνωσή της δεν υπήρχε ως στοιχείο θα υπάρξουν όλο και περισσότερε θέσει απασχόληση. Υπάρχουν και άλλε μελέτε. Την, περισσο... την περασμένη εβδομάδα, μία μελέτη έλεγε ότι μπορεί να δημιουργηθούν λιγότερε θέσει απασχόληση. Αν δείτε, α πούμε, το κόστο των ανεώσιμων πηγών ενέργεια, ε, το γεγονό ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη τι δωρεάν εκπομπέ ή τι επιπλέον εκπομπέ, είναι σαφέ ότι η μελέτη του Potsdam, του Ινστιτούτου δηλαδή Potsdam, για την ε, επίπτωση στο κλίμα ε, είναι πιο αξιόπιστη και επομένω θα έχουμε επιπλέον 6 εκατομμύρια θέσει απασχόληση. Ένα άλλο επιχείρημα είναι για την υγεία. Υπάρχουν μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής επιπλέον ε, μελέτες. Η Κομισιόν ε, είπε ότι θα μειωθεί η θνησιμότητα απλώς, αλλά οι επιπλέον μελέτες λένε ότι θα μειωθούν και οι αρρώστιες, η νοσηρότητα. Επομένως, τα ευεργετήματα για την υγεία θα είναι 36 ε, δισεκατομμύρια ε, ευρώ το χρόνο. Αν δείτε λοιπόν ε, την υγεία, τις ΕΣ απασχόλησης, τις μειωμένες εισαγωγές πετρελαίου, όλα αυτά είναι πλεονεκτήματα. Μην ξεχνάμε βεβαίως τις αναταραχές στη Βόρεια Αφρική. Υπάρχουν πάρα πολλοί οικονομικοί λόγοι λοιπόν για να θέλουμε να μειώσουμε την εξάρτησή μας από το πετρέλαιο και τις εισαγωγές πετρελαίου. Φυσικά, μετά την ακρόαση που έγραψα την έκθεσή μου, η Κομισιόν έφτιαξε αυτόν τον οδικό χάρτη, όπου λέει ότι ο στόχος του 20% ε, μέχρι το 2020 δεν είναι αποτελεσματικός σε σχέση με το κόστος. Ε. Φυσικά έχουμε επικρίσεις ε, επί της εκθέσεως της Κομισιόν και του οδικού χάρτη, ιδίως αν δείτε την καθυστερημένη δράση από πλευράς Κομισιόν και τον ισχυρισμό ότι θα έχουμε μέχρι το 2050 μείωση κατά 80%. Λέει η Κομισιόν ότι μπορούμε να ε, βασιστούμε σε αυτή την αντιστάθμιση. Εγώ πιστεύω πόση αντιστάθμιση θα υπάρξει. Νομίζω ότι οι επιστήμονες λένε ότι θα πρέπει να κάνουμε μείωση 80 με 95% και η Κομισιόν απλώς ε, συνιστά 80%. Ε, Μιλάμε για καθυστερημένη δράση Σε αυτόν τον οδικό χάρτη της Κομισιόν λέει ότι μπορούμε να έχουμε και εγχώρια μείωση κατά 25%. Ο σημερινό ευρωπαϊκό στόχο είναι 20% μέχρι το 2020 μαζί με τι αντισταθμίσει. Δηλαδή, αν φτάσετε στο 25% εγχωρίω και συμπεριλάβουμε τι αντισταθμίσει, στην πραγματικότητα φτάνουμε στο 30%. Γι' αυτό λοιπόν ζητάω ε, κάτι τέτοιο όχι εγχώρια κατά ανάγκη, παρότι υπάρχουν ε, βουλευτέ εδώ που ζητάνε εγχωρίω 30% μείωση. Και αν το ζητήσουν, εγώ δεν θα έχω κανένα πρόβλημα αυτέ τι τροπολογίε. Τέλο, για τη διαρροή του άνθρακα, το διοξείδιο του άνθρακα, που είναι βασικό στοιχείο επίση, Πρόεδρε. Ε, στο έγγραφο εργασία μου ε, κοιτάζω όλα τα επιστημονικά στοιχεία, τα ανεξάρτητα επιστημονικά στοιχεία και μελέτε, ό,τι βρήκα, εν πάση περιπτώσει, που δείχνουν ότι υπάρχει ε, περιορισμένη επίπτωση τη διαρροή του διοξίδιου του άνθρακα σε αυτή τη φάση και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα. Φυσικά γνωρίζουμε ότι αν αυξήσουμε το στόχο, η διαρροή του διοξιδίου ε, θα είναι από τα θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από αυτή την έκθεση και επομένω ε, είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη την χρηματική υποστήριξη που πρέπει να λάβουμε να βάλουμε στο περιθώριο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επενδύσουμε σε τεχνολογίες που θα μας βοηθήσουν να υλοποιήσουμε πιο φιλόδοξους κλιματικούς στόχους. Επομένως, ε, αυτά τα έσοδα από το σύστημα ανταλλαγής εκπομπών ε, τα βάζω στην άκρη. αν ε, φτάσουμε, περιοριστούμε μάλλον στο 20% μειώσει, αυτά τα έσοδα θα είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Γι' αυτό λοιπόν, αν έχουμε περισσότερες φιλοδοξίε, θα έχουμε περισσότερα έσοδα για την Ευρωπαϊκή Ένωση από το σύστημα εμπορίες ε, εκπομπών και αυτά θα τα επενδύσουμε μετά ε, σε τεχνολογίες για να αποκτήσουμε τεχνολογίε χαμηλότερων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. μαζί με την Επιτροπή Ήτρε, εκεί αυτοί έχουν ε, κάποια θέματα αποκλειστική αρμοδιότητάς τους. Ε, εγώ δεν δίνω σημασία δηλαδή στην ε, καινοτομία, στην ενεργειακή αποδοτικότητα, αλλά οι εκθέσεις της Ήτρε θα τα καλύψουν αυτά τα θέματα. Ε, αν θέλετε να βάλετε τώρα τροπολογίες για αυτά τα στοιχεία στην έκθεση, κανένα πρόβλημα. Ε, ούτως ώστε να έχουμε και εμείς ε, κάποιες απόψεις από πλευράς Επιτροπής ΕΝΔΙ και για αυτά τα θέματα. Αύριο θα γίνει επίσης ακόμα μία ακρόαση για την έκθεση για, αυτό για αυτά τα θέματα στην Επιτροπή Ήτρε. Εγώ θα συμμετάσχω και παρακαλώ και προσκαλώ τα μέλη της ΕΝΒΗ να παραστούν σε αυτή την ακρόαση της Επιτροπής Ήτρε. Πολύ ωραία. Αυτά από μέρους μου. Θα ήθελα να ακούσω τώρα τις δικές σας α, απόψεις. Ε, το χρονοδιάγραμμα είναι το ίδιο μέχρι το τέλο του Ιουνίου. Ελπίζω να έχουμε τη θέση του Κοινοβουλίου, τόσο ώστε να επηρεάσουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να δούμε αν τελικά θα αυξήσουμε τι φιλοδοξίες από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα. Εγώ λέω να αυξήσουμε αυτέ τι φιλοδοξίε. Ε, Ευχαριστώ. Μπα που μας παρουσίασε αυτή την έκθεση. Δουλεύουμε και συνεργαζόμαστε εκ του σύνεγγυς με την Επιτροπή Βιομηχανίας, την Ήτρε. Και ο εισηγητής Τη επιτροπή είτε δυστυχώ δεν είναι παρόν εδώ, αλλιώ θα του είχα δώσει το λόγο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο από του κοιόδης συζητητέ. Ο Σαλβατόρ Ταταρέλα θα πάρει πρώτο το λόγο. Ε, δεν είναι εδώ. Ποιο θα πάρει το λόγο από μέρου του ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μια ενδιαφέρουσα έκθεση του συναδέλφου μας του Μπάς. Επί της ουσίας, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η κλιματική αλλαγή, επομένως, ε, έχουμε εδώ αυτό το στόχο του 20%, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο 30% υπό τον όρο ότι θα υπάρξει διεθνή συμφωνία. Γιατί οι μεγάλε χώρε, οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Κίνα δεν θα ήταν έτοιμοι να δεχτούν μια τέτοια... Δεν είναι έτοιμοι να δεχτούν μια τέτοια συμφωνία μέχρι στιγμή. Παρότι εμεί κάνουμε προσπάθειες ε, για τη μείωση. Δεν ξέρω αν η Ευρώπη θα καταφέρει να τις πείσει και αν θα καταφέρει να πείσει, στην, ε, να πείσει τη βιομηχανία ότι μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί από ενεργειακή άποψη χωρί να δαπανούμε πολλά λεφτά για το, αυτό, το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Οι στόχοι της Κομισιόν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εδώ μιλάμε για 16 με 17%, κάτι που θα κόστιζε πολύ πιο ακριβά για... στη βιομηχανία. Για αυτό το... αυτό το λόγο ακριβώς δεν θα μπορούσαμε να δεχτούμε να περάσουμε μονομερός στο 30%. Για τη γραμμική μείωση δεν είναι να συμφωνούμε. Πιστεύουμε ότι αν καθυστερήσουμε, ε, αν είχαμε ένα διαφορετικό σύστημα εκπομπών, θα μας κόστιζε ε, λιγότερο ακριβά. Επίσης, για το θέμα της διαρροής. Ο Μπάς μίλησε γι' αυτό. Έχουμε πρόβλημα με τη διαρροή. Στην Ευρώπη θα χρειαστεί να επενδύσουμε μαζικά. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει νόημα στα πλαίσια της καταπολέμησης κλιματικής αλλαγής. Χρειάζονται τεράστιες προσπάθειες. Αυτή τη στιγμή ε, τι θα σέψουμε αυτό το πρόβλημα της διαρροής του άνθρακα, τότε μπορούμε να περάσουμε σε πιο αυστηρά μέτρα. Αλλά είναι μία εκ των όνου προϋπόθεση. Σε ό,τι αφορά τώρα την αποτελεσματικότητα, θα πρέπει να δούμε την αρμοδιότητα που έχει η Επιτροπή Ήτρε. Είναι καθήλυνα αρμόδια επιτροπή γιατί νομίζω ότι θα βαρύνει πολύ ο λογαριασμός ενέργειας. Επομένω, 20% ναι, αλλά 30% μόνο εφόσον δεχτούν και οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ, επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ τον εισηγητή, λέει ο κ. Γιώργενσεν, για την θαυμάσια έκθεση. Συμφωνώ σχεδόν με όλα τα σημεία. Θα περιοριστώ λοιπόν σε κάποια σχόλια και σε κάποιες απαντήσεις αυτά που είπε ο προηγούμενο ομιλητής και να, κάνω και κάποιες, να πω και κάποιες ιδέες, ας πούμε, για να βελτιώσουμε την έκθεση. Καταρχά το επιχείρημα ότι θα πρέπει να πάμε στο 30% μόνο εφόσον και οι άλλοι κάνουν αντίστοιχε προσπάθειες. Είναι σαν να λέμε τελικά ότι όχι, δεν θέλουμε το 30%. Τότε ας κάνουμε μία έκθεση ε, μονολεκτική που να λέει όχι. Γιατί δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Αν δούμε τις διεθνείς διαπραγματεύσει που βρίσκονται τώρα, ελπίζουμε να υπάρξει πρόοδος, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει πρόοδος, αλλά ένας από τους βασικούς εταίρους, οι Αμερικανοί, βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου μάλλον δεν θα μετακινηθούν. Και δεν θα μετακινηθούν μόνο και μόνο για να συγκριθούν μαζί μας. Η κυβέρνηση Ομπάμα έκανε προτάσεις για ένα νέο λογαριασμό για το διοξείδιο του άνθρακα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές αυτός ο, αυτό το νομοσχέδιο δεν πήγε στο Κογκρέσο αλλά όχι στην Γερουσία. Αν είχε πάει θα σήμαινε μείωση των εκπομπών κατά 16 ή 17% μέχρι το 2020. Ε, συγκρίσουμε το 2005. Εμείς ε, συγκρίνουμε το, με το 1990. Άρα ο πραγματικός, ε, το πραγματικό νούμερο στην πραγματικότητα είναι 3%. Αλλά δεν μπόρεσε να το περάσει ούτε αυτό το ελάχιστο. Και πριν Μάλιστα πριν τι ενδιάμεσε εκλογές. Άρα αποκλείεται τώρα να πλησιάσουν τους δικούς μας στόχους μείωση εκπομπών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κουνιέται τίποτα στις ΗΠΑ. Όχι. Ε, και σε επίπεδο πολιτιών γίνονται πράγματα. Ε, διάφορες εταιρείες κάνουν προσπάθειες από μόνους. Αν περιμένουμε όμως τις πολιτικές αποφάσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο, είναι σαν να λέμε ότι δεν κάνουμε τίποτα εμείς. Αν λοιπόν αυτή είναι η γνώμη κάποιων πολιτικών ομάδων εδώ στο Κοινοβούλιο, εντάξει θέμα Αλλά στο πούνε. Παρά να μας ψεματίζουν ότι πιστεύουν στη μείωση. Γιατί δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα έτσι. Τώρα, επ' αυτόν, επ' όσον λέει, εφόσον, αναφέρει έκθεση. Το πιο σημαντικό επιχείρημα είναι ότι ακόμα και αν δεν συμφωνούμε με τις φιλοδοξίες μας για μείωση των εκπομπών και για λύση στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, αν δεν θέλουμε να σώσουμε τον πλανήτη, ας δείξουμε τουλάχιστον ότι συμφωνούμε στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής οικονομίας. Είδα όλα τα στοιχεία που ανέφερε και ο Μπάς και πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι οι περιφέρειες ανά τον κόσμο και διάφορες χώρες που είναι πιο ενεργειακά αποδοτικές θα είναι και οι πιο, θα είναι και ανταγωνιστικές. Βέβαια δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιε είναι οι τεχνολογίε που θα μα κάνουν πιο αποδοτικέ, δεν ξέρουμε ποιε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια θα είναι οι πιο ανταγωνιστικέ. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό, αλλά κανένα δεν μπορεί να αρνηθεί ότι ο παλιό τρόπο παραγωγή ενέργεια και κατανάλωση ενέργεια που βασίζεται στα, ορικά στα ορυκτά καύσιμα, αυτό δεν θα είναι ανταγωνιστικό. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό. Ας δούμε λοιπόν τι πολιτικά εργαλεία θα χρησιμοποιήσουμε. Κάποια από αυτά που είπε ο Μπάς είναι καλά. Θα μπορούσαμε επίση να μιλήσουμε για ελάχιστες τιμές για τα δικαιώματα διοξιδίων του άνθρακα. Αυτό δημιουργεί κίνητρα για να υπάρξουν αλλαγέ. Επίσης, δίνει και μια βεβαιότητα στη βιομηχανία ε, για το τι να περιμένει είπες και συμφωνώ ότι πρέπει να περιμένουμε και τις άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές, κυρίως την Επιτροπή Ήτρε, αλλά το θέμα της ενεργειακής αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας συνδέεται με όλα όσα κάνουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν να μιλήσουμε για αυτό το θέμα στην έκθεση. Εγώ θα κάνω λοιπόν μια τροπολογία για αυτό το θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας. ευχαριστώ πολύ. Thank you. Uh, Ευχαριστώ. Chris Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Μπάς. Αρχικό σχέδιο ήταν ότι εμεί θα αυξάναμε το στόχο μα στο 30% είχαμε διεθνή συμφωνία. Και όταν ε, συμφωνήθηκε αυτό, Νομίζω ότι η υπόθεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ότι θα κάναμε εδώ μια γενναιόδορη χειρονομία, δηλαδή θα αναγνωρίζαμε ότι είχαμε ιστορικές ευθύνες και θα είχαμε ηγετική θέση. Νομίζω έχουν αλλάξει τώρα τα επιχειρήματα. Βλέπουμε τώρα οικονομικά επιχειρήματα όλο και περισσότερο ότι πρέπει να κάνουμε μεγάλες επενδύσεις στην τεχνολογία χαμηλών κομπομπών άνθρακα. Όπω και να έχει, πρέπει να κάνουμε επενδύσει στην παραγωγή ενέργεια και τώρα διακινδυνεύουμε να εμπλακούμε σε τεχνολογίες με ψηλές εκπομπές άνθρακα εκτός και αν κάνουμε αλλαγές. Ε, πρέπει να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι θέμα η οικονομικής επιβίωσης, γιατί αν θα είμαστε μεταξύ των πρώτων δυνάμεων παγκοσμίω ή αν θα μας ξεπεράσουν ε, αναδυόμενες οικονομίες. Ε, και είναι αναφυσβήτητο ότι τώρα πρέπει να αλλάξουμε ταχύτητα. Αυτό βέβαια δεν ε, έχει αναγνωριστεί ακόμα από πολλά μέλη από αυτό το κοινοβούλιο και ούτε το έχει αναγνωρίσει και το Συμβούλιο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ε, ο συνάδελφος στο Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται να είναι μεταξύ των ε, ε, υποστηρικτών που προσπαθεί να αυξήσει το στόχο στο 30% μεταξύ του Συμβουλίου. Ο Κρίς ήταν για έξι χρόνια μέλος αυτού του Κοινοβουλίου και πάντα δεν ήταν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, αλλά χαίρομαι τελικά που αναλαμβάνει τώρα αυτή τη δράση. Την περασμένη εβδομάδα ακούσαμε την Κομισιόν να, ε, να ανακοινώνει τον οδικό της χάρτη για οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ο αρμόδιος επίτροπος για την κλιματική αλλαγή είπε ότι οι απαιτήσει για αυτό τον οδικό χάρτη είναι να αυξήσουμε το στόχο μας τουλάχιστον στο 25% μέχρι το 2020. Όμως, ε, από ό,τι φαίνεται, δεν λαμβάνει την απαραίτητη υποστήριξη από την Κομισιόν. Παραγωνίζεται για να θέσει αυτούς τις απαιτήσει και τους στόχους. Έτσι λοιπόν, τώρα οπισθοχωρεί και επανέρχεται στον ισχυρισμό ότι αν εφαρμόσουμε όλη την νομοθεσία ε, που υπάρχει ήδη πλήρως, τότε θα φτάσουμε στο στόχο του 25%. Ναι. Ίσως. Αλλά επίσης η Επίτροπος δηλώνει ότι σήμερα έχουν μειωθεί οι εκπομπέ μα ε, κατά 17% σύμφωνα με την επίπεδο του 1990. Και φαίνεται να είμαστε μακριά το 17 μέχρι το 25 ή παραπάνω, αλλά λάβατε και την επιστολή από την Ζακλίν Μαλέκ από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος που είπε ότι το 1 τρίτο των μειώσεων που έχουν επιτευχθεί είναι αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης τα τελευταία δύο έτη. Έτσι, λοιπόν, εδώ μιλάμε για κάτι πολύ ευρύτερο από αυτό που είπε η Επίτροπος. Εδώ 13% μείωση σε σχέση με το επίπεδο των 90%. Και έχουμε και το θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας. Στόχος 20% μέχρι το 2020. Σίγουρα δεν θα μας ε, οδηγήσει στο να βελτιώσουμε την ενεργειακή μας αποδοτικότητα παρά μόνο κατά 9% μέχρι το 2020 ο Επίτροπο ενέργεια είπε ότι είναι έτοιμο να παρουσιάσει υποχρεωτική νομοθεσία αλλά πρέπει να πιστεί πρώτα, να είναι πεπισμένο ότι θα σεβαστούν τα κράτη-μέλη του στόχου. Έτσι λοιπόν όλα αυτά δεν θα ε, παρουσιαστούν μέχρι το 2013 και αυτό σημαίνει ότι δεν θα τεθούν σε εφαρμογή μέχρι το 2015. Ε, βλέπουμε ότι δεν είναι και τόσο δυναμική η επίδοση της ε, Κομισιόν. Ε, Επίτροπος λέει ότι πρέπει να έχουμε μία τιμή για τον άνθρακα προκειμένου να προωθήσουμε τις επενδύσεις για τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα. Δεν μπορεί βέβαια να δει επίτροπο πώς ε, οι κυβερνήσεις και οι Κομισιόν θα υποστηρίξουν ε, μια μείωση του ανώτατου ορίου. Έτσι λοιπόν πιστεύει ότι είναι δυνατόν ε, να μην ετεθούν σε εμπορία κάποια από τα δικαιώματα που έχουν στη διάθεσή του οι κυβερνήσει. Όμως τι θα γίνει, θα αυξηθεί η τιμή ακόμη και στα 20 ευρώ ανατόνο. Ορισμένοι λένε ότι χρειαζόμαστε 30 ευρώ ανατόνο για να γίνουν οι απαραίτητες επενδύσει. Δεν έχω δει καμία δήλωση όμω από την Κομισιόν. Ίσως υπέθεσταν ότι θα υπάρχει τόσο ταχύ οικονομική ανάπτυξη τα επόμενα έτη που η τιμή θα αυξανόταν επειδή θα αυξανόταν και ζήτηση. Όμως να δω κάτι από την Επιτροπή σε σχέση με τις προβλέψεις. Όλα όλα αυτά δεν τα λέω μόνο εγώ. Η ε, Euroelectric που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Μηχανή Ελεκτρισμού έχει το δικό της οδικό χάρτη για να πετύχει παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με μηδενική παραγωγή εκπομπών ε, μέχρι το 2050 και λέει ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό με τα μέσα που υπάρχουν τώρα. Είναι πάρα πολύ χαμηλή η τιμή του άνθρακα. Έχουν γίνει κάποιες επενδύσεις που είναι ελκυστικές για τις εταιρείε για να λάβουν, παραδείγματος χάρη, επιδοτήσεις από τις κυβερνήσεις ε, για ένα project ολικής ενέργειας, αλλά δεν ε, μιλάμε για λογικές επενδύσεις σε πολλές ε, περιπτώσεις. Έχουμε πάρα πολλά φωτοβολταϊκά στη Γερμανία και στην Βόρεια Ευρώπη. Δεν χρησιμοποιούμε όρθα τα χρήματα με τον τρόπο αυτό. Και να πω και κάτι άλλο. Αν δούμε τις οικονομικές προβλέψεις, η Κομισιόν βασίζει την περισσότερη δουλειά της σήμερα σε εκτιμήσεις για την τιμή του πετρελαίου για 105 δολάρια μέχρι το 2020. Όλες οι δικές μας υποθέσεις βασίζονται λοιπόν σε αυτή τη τιμή. Τώρα δεν ξέρω, έχουμε 137, είναι η τιμή ε, του πετρελαίου. Είναι πολύ υψηλότερη και ίσως να μην ξανακατεύει. Είδαμε και τις ε, εκθέσει που ήρθαν από το Γερμανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τονίζεται η ανάγκη για αυξημένε επενδύσεις. Αν αυξήσουμε το στόχο αυτό ε, από το 20 στο 30 θα δώσουμε όθηση στην οικονομία μας. Ε, θα έχουμε περισσότερες επενδύσεις και θα είμαστε σε καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσουμε την ανάπτυξη τη κινέζικης οικονομία και των οικονομιών της από Διαφορετικά δεν θα προωθηθεί η, η ευρωπαϊκή οικονομία. Έτσι λοιπόν πρέπει να προωθήσουμε αυτά τα οικονομικά επιχειρήματα επίση για την αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ και τον συνσηγητή τον κύριο Κρίς Ντέιβις. Όμως θα ήθελα να ζητήσω από τους υπόλοιπους συνεισηγητές να μην μακρηγορήσουν τόσο πολύ, διαφορετικά δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Μύροσλαβ. Ευχαριστώ. Θα δράξω αυτή την ευκαιρία για να μιλήσω τσεχικά. Ακούσαμε πολλά επιχειρήματα με τα οποία μπορώ να συμφωνήσω. Θα ήθελα να σας εξηγήσω γιατί τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Αν και κατανοώ την αξία του έργου του συζητητή. Δεν βλέπω μία αναφορά στο μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στις παγκόσμιες εκπομπές, δηλαδή πώς εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε και τι μπορούν να κάνουν οι άλλες χώρες. Αναφέρθηκαν οι Ηνωμένε Πολιτείε από τον συνάδελφο. Τι μπορούν να κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε για να μειώσουν τις εκπομπές. Αν ε, είχαν υιοθετήσει την απαραίτητη νομοθεσία. Βέβαια, ενοχλούμε πάρα πολύ όταν ακούω και το άκουσα και στον Ελλομέλιο ότι πρέπει να είμαστε επιφιλόδοξοι, γιατί η Κίνα έχει συμφωνήσει σε μείωση 40% μέχρι το 2020. Ελπίζω όλοι σε αυτήν την επιτροπή να γνωρίζουν ε, ότι εδώ συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Η Κίνα υποσχέθηκε να μειώσει τη σχεδιαζόμενη αύξησή της, που ήταν 200%. Δηλαδή θα μειώσουν αυτή την προβλεπόμενη αύξηση κατά 40%. Δηλαδή το 2020 η συνεισφορά των Κινέζων στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής θα είναι συν 160%. Ω προ τι εκπομπέ. Έτσι λοιπόν, αν στην Ευρώπη μειώσουμε τι εκπομπέ και 100%, δεν θα έχει αυτό αποτέλεσμα στην κλιματική αλλαγή, γιατί ο υπόλοιπο κόσμο δεν θα συνεργάζεται. Εγώ παρευρέθησα στις τελευταίες τέσσερις διασκέψεις για την κλιματική αλλαγή. Ήμασταν και με την ελπίδα ότι θα υπήρξε ένα συμβιβασμό, μπορούσαμε να μιλήσουμε στι αναπτυσσόμενε χώρε, στι αναπτυσσόμενε οικονομίε. Τελικά ξέρουμε ότι τίποτα δεν προέκυψε. Έτσι λοιπόν Εμεί μπορεί να είμαστε φιλόδοξοι ως προς μας αλλά δεν θα πετύχουμε τίποτα. Μπορούμε να πετύχουμε κάτι μόνο ε, σε επίπεδο οικονομικών κινήτρων. Στην Ευρώπη θα πρέπει να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα. Θα έπρεπε να προωθήσουμε, να δώσουμε όθηση στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, όμω δεν το κάνουμε και πολύ καλά αυτό. Εδώ και 6 χρόνια ακούω πώ θα αυξηθούν θέσει εργασία στην Ευρώπη με τι νέε τεχνολογίε. Όμω αυτό που βλέπουμε είναι ότι η ενεργία αυξάνεται στην Ευρώπη. Ε, διοικητικά μέτρα για την προώθηση τη ενέργεια από νέε πηγέ έχουν οδηγήσει μόνο σε αύξηση 20% στις ε, τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τις επιχειρήσεις και 14% για τα νοικοκυριά. Ως αποτέλεσμα της παραγωγής ε, ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιακή ενέργεια. Δεν νομίζω ότι αυτό ήταν λογικό το σχέδιο. Αυτό το σχέδιο ήταν λογικό, με συγχωρείτε. Έτσι όπως ε, το είχαμε σχεδιάσει τη στιγμή λήψη της απόφασης. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να λέμε κάτι στην έκθεση και για τη διεθνή συνεργασία. Θα πρέπει να λέμε και τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη σε ρεαλιστικό επίπεδο. Γιατί όλες αυτές οι αποκαλούμενες ανεξάρτητες μελέτες σύμφωνα με τις οποίες ε, μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα θα μας ε, οδηγήσει στην παγκόσμια οικονομική ε, είναι κάτι που υπάρχει μόνο στο χαρτί, είναι κάτι θεωρητικό. Ξέρουμε ότι μετεγκαθίστανται οι βιομηχανίες από την Ευρώπη, ότι η Ευρώπη χάνει εναντί λοιπόν χωρών ως προς τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Έτσι λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις εκπομπές μας και την ε, εξάρτησή μα από τα ορυκτά καύσιμα, αλλά μην δώσουμε τη χαριστική βολή στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αυτό Τι είναι αυτό, πολωνικά ή τσέχικα. Σας ευχαριστώ πολύ, στα τσέχικα. Η τσεχικα σα ευχαριστω πολυ στα Βίλτσα. Α, δεν είναι εδώ. Ρώση. Ευχαριστώ. Βρισκόμαστε στο γνωστή δέσμη μέτρων για το κλίμα, μάλλον ίσως ε, θα από ό,τι φαίνεται κάποιοι σκέφτονται ότι οι σεισμοί προκαλούνται από τις κλιματικές ε, αλλαγές. Ε, κάποιοι σκέφτονται ότι η γη δεν είναι στρογγυλή και κάποιοι πιστεύουν ότι αν μειώσουμε τις εκπομπές 30% μέχρι το 2020 θα έχουμε περισσότερες ε, θέσεις εργασίας. Έλεος. Ε, το θέμα είναι ότι βρισκόμαστε τώρα στο 20% και θα μπορούσαμε να είμαστε και πιο πάνω, γιατί πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουν κλείσει ή μεταγκαταστάθηκαν λόγω της κρίσης και δεν νομίζω ότι αυτό δημιουργήσει ένα αίσθηση εργασίας. Το αντίθετο, το ποσοστό των ανέργων έχει αυξηθεί σήμερα στην Ευρώπη. Όμως ε, φυσικά πιστεύω ότι ο εισηγητής πιστεύει αυτά που λέει τουλάχιστον. Ωραία, είδαμε ότι αναφέρεται συνέχεια κάποιες μελέτες σύμφωνα με τις οποίες ότι αν αυξήσουμε, ε, μάλλον ε, αν μειώσουμε τις εκπομπές αυξάνονται οι θέσεις εργασίας και δεν υπάρχουν προβλήματα για την οικονομία. Όμως υπάρχουν και μία σειρά μελετών που λένε ακριβώς το αντίθετο. Μάλιστα εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μας εξηγείτε πως ε, μία επιχείρηση που μολύνει εδώ και που οδηγείται στο κλείσιμο γιατί δεν σέβεται τους κανόνες που εμείς θα επιβάλλουμε, αν ε, κατασταθεί σε μία τρίτη χώρα και παράγει ακριβώς τα ίδια προϊόντα, ε, και χωρίς καν ε, να περιορίζεται στο 20% για τις εκπομπές ούτε καν στο 30%. Δηλαδή, αν πάει και στην Κίνα μπορεί 160% περισσότερο να μολύνει και πρέπει να μου εξηγήσετε πώς ακριβώς αιτιολογείται σε παγκόσμιο επίπεδο ότι βελτιώνεται ε, οι συνθήκε για το περιβάλλον. Εμεί κλείσουμε μια επιχείρηση στη δική μα χώρα στην Ευρώπη, γιατί επιβάλλουμε πάρα πολλά. Αυτή θα μεταγκατασταθεί και μπορεί να εγκατασταθεί κάπου που μολύνει 160% περισσότερο. Πώ δηλαδή για το παγκόσμιο περιβάλλον. Και εγώ νομίζω το πιο παγκόσμιο που υπάρχει είναι το περιβάλλον. Δηλαδή, είτε ε, έχω εκπομπέ στην Κίνα ή στι ΗΠΑ ή στην Ελβετία, είναι κάτι παγκόσμιο. Πρέπει λοιπόν να μου εξηγήσετε πώ το ότι χορηγείται από ε, χημική σκοπιά. Δηλαδή ε, δεν ε, κάνουν κακό οι εκπομπές, ε, αν εκπέμπονται στην Κίνα, ενώ αν εκπέμπονται στην Ιταλία, κάνουν κακό και μας ε, σκοτώνουν κιόλα. Και ακούσαμε τι είπε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ε, δαπανηρές μελέτες, ενώ η Επιτροπή μας είπε ότι μέχρι το 2020 θέλει να διπλασιάσει την παραγωγή της ενέργειας και θα διατηρήσει απαράλλαχτα τα ποσοστά για τις ε, εναλλακτικέ πηγές ε, ενέργειας ε, αλλά και για την παραγωγή ενέργειας. Μπορείτε να μας πείτε πόσοι μελέτες λένε ότι αν μειώσουμε τις εκπομπές θα είναι καλύτερη η κατάσταση μόνο την Ευρώπη αλλά δεν μιλάτε για την Κίνα αναλόγως πολλές φορές το κόκκινο πάει με το πράσινο αλλά πρέπει να μας τα εξηγήσετε αυτά. Ίσως να φτάσουμε στο 17% για το 2020, αλλά σε σύγκριση με το 2000. Προσοχή, όχι σε σχέση με το 1990 όπως θέλουμε να κάνουμε εμείς και πρέπει να μου εξηγήσετε και ένα άλλο χημικό θαύμα γιατί η Επιτροπή στη σελίδα 11 Τη έκθεση λέει ότι αν δεν κατορθώσουμε να μειώσουμε κατά 3% τι εκπέσει διοξιδίου του άνθρακα, τότε ε, θα ε, έχουμε και ε, λιγότερα εργαλεία για να μειώσουμε άλλες ε, άλλες ουσίες όπως πρέπει να τους χάσει ουσίες προκύπτουν από τα βαρέα μέταλλα. Έτσι λοιπόν πρέπει να μου πείτε αν ε, το 30% ε, μείωση σημαίνει ότι θα κλείσουμε τις χι επιχειρήσεις και επομένω θα μειωθούν και περαιτέρω οι εκπομπές. Όμως από χημική σκοπιά πώς μπορείτε να μου εξηγήσετε ότι αν μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα μειώνουμε και τις εκπομπές από τα βαρέα μέταλλα στην ατμόσφαιρα. Άλλο σημαντικό θέμα και θα φτάσω τώρα και σε αυτό το θέμα της υγείας. Ο εισηγητής αναφέρεται στο εξή ότι υπάρχουν ε, ε, και αυτά τα ωφέλη για την υγεία. Μπορώ να σας πω το εξή. Αν άλλες χώρες συνεχίζουν να μολύνουν ακόμη περισσότερο και το έδωσε ε, το παράδειγμα συνάδελφος από το ΕΣΥΑΡ, δηλαδή αν ακόμη και εμείς σβήναμε την Ευρώπη και συνέχιζε η Κίνα την πορεία που έχει εξαγγείλει τότε αν ε, δεχτούμε ότι θα σβήσουμε την Ευρώπη, ούτε ένα καυστήρα, δεν θα χρησιμοποιούμε τίποτα. Έτσι λοιπόν εξαφανίζεται η Ευρώπη, η Κίνα κάνει αυτό που έχει εξαγγείλει. Έτσι λοιπόν πρέπει να μου εξηγήσετε πώς είναι δυνατόν να φανταστούμε καταστάσεις ε, που ε, θα είναι καλύτερε από τη σκοπιά τη υγεία, που θα βελτιώσουν την υγεία. Αν γνωρίσουμε ότι ακόμη και αν σβήσουμε την Ευρώπη μόνο χάρη στην Κίνα, θα έχουμε περισσότερες μολυσματικές ουσίες. Δηλαδή θέλω να μου, μου εξηγήσετε πώς είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και εγώ σαν μέλος της Επιτροπής έχω βάλει το όνομά μου στον κατάλογο. Εδώ μιλάμε για την πρόταση όσον αφορά τα ποσοστά πέρα των 20% μείωση. Και μιλάμε βέβαια για το 2020, τους στόχους που έχουν θέθει. Η όλη συζήτηση λοιπόν που κάνουμε τώρα θα πρέπει ίσως να μπει σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή να κινηθούμε αν θέλετε σε έναν άλλο προσανατολισμό. Να δούμε το οικονομικό μοντέλο το οποίο θα βασίζεται σε μια δραστηριότητα με λιγότερο άνθρακα. Και το ερώτημα είναι αν αυτή η πρόκληση μπορεί να μετατραπεί σε μια ευκαιρία για την Ευρώπη. Και όταν μιλάμε για την ανεργία, για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, διαπιστώνουμε ότι οι επενδύσεις που πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να έχουν σαν αποτέλεσμα εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και μεταβολή των συστημάτων των πηγών ενέργειας και αυτό μπορεί να είναι όντως μια ευκαιρία για περιοχές της Ευρώπης που δεν έχουν παράδοση σε βιομηχανική παραγωγή ή τουλάχιστον δεν έχουν μεγάλη παράδοση. Για αυτές τις περιοχές θα μπορούσε το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος, της οικολογίας να ειδωθεί και από την άποψη της βιομηχανικής πολιτικής. Και να υπάρξει ένας ανταγωνισμός μεταξύ Ασίας, Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας μέσω των νέων τεχνολογιών και των εφαρμογών. Αυτό είναι το θέμα που μας αφορά. Το 20 ή 30% αν θέλετε είναι συμβολικές αξίες. Θέλουμε δηλαδή να προχωρήσουμε, να εξελιχθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και είναι ενδεικτικά θα έλεγα αυτά τα ποσοστά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ε, να μην κοιτάμε μόνο το οικολογικό, το περιβαλλοντολογικό κομμάτι, την προστασία του περιβάλλοντος και την, το κλίμα, αλλά και την οικονομική συνιστόσα. Να δούμε δηλαδή οι νέες επενδύσεις σε τι οδηγούν και να τις κατευθύνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Άκουσα τον ωραίο στο Ρώση με προσοχή αυτά που είπε για την βιομηχανία, την Κίνα το πακέτο για το κλίμα και βεβαίως το σύστημα συναλλαγής ε, εκπομπών και ποιος είναι ο στόχος μας εκεί. Έχουμε αυτό το 60% εκτός του πακέτου του συστήματος ε, συναλλαγών. Και βεβαίως υπάρχουν δυνατότητες εδώ να κινηθούμε προς μια καλύτερη αντιμετώπιση. Η ερώτηση είναι τώρα. Η απόφαση που λαμβάνουμε, που έχει στρατηγική σημασία, που λαμβάνει εδώ η Επιτροπή Περιβάλλοντος, για αυτό το 20%, στέλνεται με αυτή την απόφαση ένα μήνυμα προς ε, αυτούς που ενδιαφέρονται, προς την κοινή γνώμη, προς τους φορείς και εδώ στην Επιτροπή μας, Επιτροπή ΕΜΒΗ, αλλά και στην Ολομέλεια, έχουμε πει ότι πρέπει να είμαστε στην πρωτοπορία. Γι' αυτό και μιλήσαμε για το 30%. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να το σκεφτούμε αυτό και να το κάνουμε. Δεν μπορεί η Επιτροπή Περιβάλλοντος να υποχωρήσει και να επανέλθει στο 20%. Δεν είναι δυνατόν να υποχωρήσουμε και να πούμε «Όχι, κάναμε λάθος, θα παραμείνουμε στο 20% και όλα τα άλλα είναι πολύ φιλόδοξα, ας τα ξεχάσουμε». Στο το 2011 στο 17,3%. Εγώ χτες ήμουν εδώ σε ένα δείπνο με συζήτηση για τα εθνικά σχέδια όσον αφορά τις ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας. Και τα ποσοστά που ακούστηκαν είναι 20-21% και πολύ περισσότερο. Αυξάνεται το ποσοστό δηλαδή της ενέργειας που παράγεται από τις ε, νέες αυτές πηγές ενέργειας. Νομίζω λοιπόν ότι θα το καταφέρουμε χωρίς να υπάρξει μεγάλη μεταφορά της βιομηχανικής παραγωγής στην Κίνα. Πρέπει ο εξυγχρονισμός να ακολουθεί και την οικονομική πολιτική. Ήθελα και εγώ να εκφράσω τις απόψεις μου. Ο Πίτερ Λίζα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ γιατί κανείς εδώ σε αυτή την Επιτροπή δεν έχει αμφισβητήσει τους μέχρι τώρα ε, στόχους που έχουμε θέσει. Ε, δυστυχώς είδατε τι συνέβη στην Ιαπωνία και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και που δεν είναι λόγο να μην μειώσουμε τους στόχους μας, τα πρότυπά μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα ε, της αλλαγής του κλίματος θα πρέπει να συνεχίσουμε να το παίρνουμε πάρα πολύ στα σοβαρά. Η καταστροφή στην Ιαπωνία είναι κάτι που σίγουρα θα μας απασχολήσει. Πολλοί θα αλλάξουν την απόψή τους όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια, αλλά είναι καθοριστικό το θέμα της αλλαγής του κλίματος. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι κάτι σημαντικό. Η αποτελεσματικότητα και η απόδοση της ενέργειας, όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε συνδυασμένα και σήμερα στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που σαφώς μας καλούν να δώσουμε κάποιες απαντήσεις. Απαντήσεις ε, που μας οδηγούν ε, προς τα μπρος. Τώρα, όσον αφορά αυτό το 20% ή 30%. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή στην ε, Επιτροπή. Είμαστε ένα σοβαρό όργανο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν όμως πολλοί φορείς και στα κρατημέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν πάρει αποφάσεις. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να παραμείνουμε στυλωμένοι στις αρχικές μας θέσεις. Δεν μπορεί να είναι αυτή η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν τρεις ε, υπουργοί της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας, Υπουργοί Περιβάλλοντος, έχουν μιλήσει για αυτό το 30%, το έχουν στηρίξει, δεν υποστηρίζονται βέβαια ακόμα από τις κυβερνήσεις τους. Οι στόχοι πάντως είναι γνωστοί και όντως υπάρχει για πολλά όργανα, για πολλούς θεσμούς εδώ μία διαμάχη. Μπορούμε βεβαίως να παραμείνουμε επί τρία χρόνια σε αυτή την κατάσταση. Ο ένας να λέει 20% και ο άλλος 30%. Όμως όμως πιστεύω ότι πρέπει να βρεθούμε σε μια διαφορετική κατάσταση και να κάνουμε έναν συμβιασμό. Η πρότασή μου λοιπόν για συμβιβασμό είναι η εξή. Να πάμε από το 20% στο 25% και να πούμε ότι αν γίνουν προσπάθειες με αποτέλεσμα σε πολλά κράτη-μέλη τα επόμενα χρόνια να συνεχίσει να υπάρχει επί ε, η πρόταση για το 30% να ανοίξουμε δηλαδή το 25% σαν ένα πρώτο βήμα και να πούμε ότι από εδώ και πέρα θα εξετάσουμε προσεκτικά τις εξελίξεις και την πρόοδο για να δούμε αν ρεαλιστικά μπορούμε να προχωρήσουμε στο 30%. Δεν είναι μόνη της η Ευρώπη. Διαφωνώ με αυτούς που λένε το 2007, αν θυμάστε, όταν ε, τέθηκαν για πρώτη φορά αυτοί οι στόχοι για το κλίμα, είχε πολύ διαφορετική προσέγγιση από σήμερα. Θυμάστε παραδείγματος χάρη η Βραζιλία, η πέμπτη οικονομία όσον αφορά το θέμα που μας αφορά. Είχε πει ότι μειώνοντας κατά 29-30%, 33% τις εκπομπές της και μιλάμε εδώ για μια χώρα που γνωρίζεται την κατάσταση της οικονομίας της. Το Μεξικό 30%. Τώρα με την Κίνα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Ξέρετε ότι υπάρχουν όμως δυνατότητες τους επόμενους μήνες μέσω των διαπραγματεύσεων να συμπεριφερθεί λίγο πιο επικοδομητικά, λίγο πιο θετικά. Δεν είμαστε όμως εκεί που θέλουμε να είμαστε. Δεν θέλουμε να αποδυναμώσουμε τις θέσεις των άλλων. Θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το 30%. Αυτό το 17% το οποίο ακούστηκε πλησιάζει το 20%. Ίσως λοιπόν με νέα στοιχεία πλησιάσουμε πιο πολύ. Να φτάσουμε δηλαδή το 20% και λίγο παραπάνω Πιστεύω ότι η κατάσταση δικαιολογεί μια πιο αισιόδοξη προσέγγιση. Τελειώνω. Μιλήσατε για την ανεργία. Είπατε ότι στην ανεργία αυξάνεται στη Γερμανία. Κάνουμε πολλά σφάλματα. Δεν είναι όλα τέλεια στη Γερμανία. Αλλά τουλάχιστον όσον αφορά την ανεργία είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Από τη στιγμή λοιπόν που η Επιτροπή προτείνει εδώ το 25% με μακροπρόθεσμους ε, στόχους και προοπτικές, χωρίς να αλλάξει τίποτα στο σύστημα ε, εμπορίας εκπομπών. Ας εξετάσουμε τα στοιχεία που μας δίνει εδώ η Επιτροπή. Ας δεχτούμε αυτή την πρόταση της Επιτροπής για 25% και με έξυπνο τρόπο να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη, τη διεθνή οικονομία για να δούμε πότε και πώς μπορούμε να προτείνουμε το 30 και να φτάσουμε στο 30. Πρόεδρος, ωραία. Πίτερ Λίζε, δεν είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Ανταλλάσσουμε απόψεις, ακόμα και δεν συμφωνούμε. Θα ήθελα εδώ να χαιρετήσω ένα πρώην μέλος της Επιτροπής, τον κύριο Τιουκε Άισμα, από την Ολλανδία. Από το 1994 ήσασταν μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, είστε εδώ με μια αντιπροσωπεία της αεροπορίας από την Ολλανδία. Καλωσορίσατε και είδατε τι σοβαρά θέματα συζητάμε στρατηγική στον τομέα της αλλαγής του κλίματος. Έχουμε επίσης και μια ομάδα της Κοντάντσε Κρέλ, οι οποίοι παρακολουθούν την συνεδρίασή μας. Ο Βιτόριο Πρόντι έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μπερδευτεί λιγάκι από τη συζήτηση. Γιατί βάζουμε στο ίδιο καλάθι θέματα τα οποία έχουν τελείως διαφορετική λογική. Εδώ συζητάμε τη σκοπιμότητα του να περάσουμε από το 20% στο 30% της μείωσης των εκπομπών. Αλλά το πλαίσιο αναφοράς είναι αυτό το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Προσπαθούμε λοιπόν να φτάσουμε σε μια διεθνή συμφωνία για τον έλεγχο των εκπομπών. Και ή δυνατόν να είναι δεσμευτική αυτή η συμφωνία. Η Κομισιόν κάνει αυτή την πρόταση για μια εταιρεία η οποία θα απελευθερώνεται από το, συγγνώμη, για μια κοινωνία που θα απελευθερώνεται από το διοξίδιο του άνθρακα μέχρι το 2050. Δηλαδή μιλάμε για μια μείωση 80-90% των εκπομπών. Η διαφορά τώρα σε σχέση με αυτό το έγγραφο είναι ότι η Κομισιόν λέει ότι αυτό μπορεί να γίνει ούτως ή άλλως, γιατί βολεύει, γιατί θα πληρώνουμε λιγότερο τα ορυκτά καύσιμα, γιατί θα υπάρχουν ε, ευεργετήματα ευεργετήματα για την υγεία, ευεργετήματα για το περιβάλλον κτλ. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε ανεξάρτητα από άλλους να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο για μια κοινωνία χαμηλού άνθρακα, χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Και επομένως έτσι αλλάζουμε και τη γενικότερη φιλοσοφία μας. Αν μπορούμε να προχωρήσουμε μόνοι μας, τότε, τότε μπορούμε να σκεφτούμε τελείως διαφορετικά το θέμα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Δηλαδή, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι τρόποι διαφορετικοί από το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Παραδείγματο χάρη ένας φόρος για την εκπομπή του διοξιδίου του άνθρακα, με μία αντιστάθμιση στα σύνορα, στο τελωνίο, για εκείνους που εκπέμπουν τελικά διοξείδιο του άνθρακα και που δεν σέβονται την πειθαρχία που εμείς ε, ή τα μέτρα που εμείς υιοθετούμε. Πριν προχωρήσουμε στη συζήτηση, θα πρέπει να καταλάβουμε λίγο το σενάριο και για αυτό το ενδεχόμενο του περάσματος από το 20% στο 30% ή και παραπάνω της μείωσης των εκπομπών. Θεωρώ και το λέω και στον εισηγητή ότι θα ήταν ενδιαφέρον να συζητήσουμε εάν μπορούμε μαζί με την Κομισιόν να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποια είναι η λογική που πρέπει να ακολουθήσουμε. Και Εν τη αυτή περιπτώσει ε, θα πρέπει να έχουμε μια συμπεριφορά από σήμερα μέχρι το 2050 ε, συνεπή. Ε, πιστεύω ότι αυτές οι δύο λογικές μπορεί να είναι αντιφατικές, γιατί είναι ε, συμπληρωματικές λογικές, διαφορετικές και σε ό,τι αφορά την παραγωγή της ενέργειας και σε ό,τι αφορά το γενικό τρόπο που ρυθμίζουμε το, την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το σκεφτούμε πριν κάνουμε οποιαδήποτε άλλη συζήτηση. Ευχαριστώ grazie. Corinne Lepage. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, υπόθηκαν πολλά πράγματα, αλλά θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο Πίτερ Λίζε, κυρίως. Ε, Βεβαίω, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να περάσουμε στο 30% και ίσως και παραπάνω. Αυτά που ζούμε, αυτά που συνέβησαν στην Ιαπωνία, ε, ξαναμοιράζουν τα χαρτιά στον ενεργειακό τομέα. Τίποτε θα είναι όπως το ζήσαμε μέχρι τώρα, μετά από αυτά που συνέβησαν στην Ιαπωνία. Ούτε σε ό,τι αφορά την πυρηνική βιομηχανία, ούτε σε ό,τι αφορά την ευαισθησία του πλανήτη στα περιβαλλοντικά και κλιματικά θέματα. Είτε για το θέμα τη πυρηνική ενέργεια, είτε για το θέμα τη κλιματική αλλαγή. η αντίληψη είναι διαφορετική. Αυτό δείχνει ότι ολόκληρη η ανθρωπότητα μετά από αυτό το δράμα θα καταλάβει ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα κλιματικά θέματα γιατί είναι θέματα ζωής και θανάτου τα λέω όλα αυτά για να σας πω ότι για όλους όσους επιθυμούν ένα σύστημα ανάπτυξης όπου οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η πράσινη οικονομία ε, είναι κεντρική σημασίας, ε, που επιτρέπουν να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, όπως είπε και ο εισηγητής, για όλους αυτούς υπάρχει ένα βήμα για να ακουστούν. Και θα ήταν ε, τρελό να μην τους ακούσουμε. Αντίθετα από αυτά που ακούσαμε στην Ήτρε χθε, νομίζω ότι η στιγμή είναι κατάλληλη, η πλέον ενδεδειγμένη για να πούμε ότι είναι και η ώρα επιτέλου, για να βάλουμε όλες μας τις επενδύσεις σε αυτή τη νέα τεχνολογία, σε αυτές τις νέες τεχνολογίες, γιατί έτσι θα επιλύσουμε ταυτόχρονα και τα προβλήματα εξόδου από την παραγωγή ενέργειας από πυρηνικά μέσα, να βγούμε, να απαλλαγούμε από το πετρέλαιο, γιατί πρέπει να το κάνουμε, και το θέμα της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσης απασχόλησης. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Νομίζω ότι πραγματικά έφτασε η στιγμή για να δοθούμε ολοκληρωτικά ε, σε αυτή την ατραπό και εμείς η Επιτροπή Περιβάλλοντος, ε, Πρόεδρε, είμαστε σε θέση να το κάνουμε, να αφιερωθούμε σε αυτό το δρόμο, ε, γιατί όλοι μας οι συμπολίτες θα δεχτούν και θα ζητήσουν κάτι τέτοιο. Όλοι χρειαζόμαστε την ελπίδα και νομίζω ότι πρέπει να πιστέψουμε από, την, από το αδιέξοδο. Και με, αυτόν αυτό το δρόμο νομίζω θα το, θα το καταφέρουμε. Ο Καρλ, ευχαριστώ. Σάιτερ. Νομίζω ότι δείξατε και αυτοσυγκράτηση και θέληση για συμβιβασμό στην αρχική σας θέληση. Γιατί εσείς και εγώ και διάφοροι άλλοι πράσινοι θα θέλαμε μια εγχώρια μείωση των εκπομπών 40%. Είναι η μόνη λύση που μας δίνει μια μικρή ελπίδα για να επιτύχουμε τους κλιματικούς στόχους που έχουμε όλοι. Το καλό με αυτούς τους στόχους είναι ότι θα επιλύσει παράλληλα και το θέμα των στόχων κοινοτομίας. Όλοι θέλουμε περισσότερη κοινοτομία. Βάλτε ένα στόχο 40% τη μείωση και δείτε τι θα γίνει με την κοινοτομία. Θα φτάσουμε, θα φτάσουμε του στόχου τη κοινοτομία. Όλοι ανησυχούν για τι θέσει απασχόληση. Για σκεφτείτε ότι αν θέλουμε να φτάσουμε τον στόχο για δημιουργία θέσεων απασχόλησης, χρησιμοποιώντας την ανάπτυξη ως εργαλείο και θέλουμε να πετύχουμε το στόχο της μείωσης για τις εκπομπές, τότε θέλουμε ανάπτυξη 3-4% και θέλουμε 2-3-4% ε, μείωση των εκπομπών κάθε χρόνο. Αυτό θα μας δώσει μια αποτελεσματικότητα των ε, πόρων, ε, μια αύξηση της αποτελεσματικότητας 4-5-6% από την τελευταία έκθεση της Κομισιόν για το στόχο ενεργειακής αποδοτικότητας θα έχουμε μόνο ε, ένα στόχο 10% σε 10 χρόνια ή 15% ενεργειακή αποδοτικότητα αν είμαστε τυχεροί. Επομένως, μην ξεχνάμε ότι εδώ δεν φτιάχνουμε μια γνωμοδότηση για αυτή την για τα θέματα που έχουμε αρμοδιότητα, μάλλον που έχει αρμοδιότητα η Επιτροπή Ήτρε. Ε, δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχουμε και τους στόχους ε, της ανεργίας, ούτε και τους στόχους της μείωσης, ούτε το 20% ούτε το 30%. Εκτός και αν εξοικονομήσουμε ενέργεια και αυτό γίνει υποχρεωτικά. Και αυτό θα είναι το πιο αποτελεσματικό ε, σε σχέση με, το κόστος για να βρεθεί λύση και στην κλιματική κρίση, ε, πρόβλημα με την πυρηνική ενέργεια και τα δικτά καύσιμα. Χρειαζόμαστε ε, επομένως μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας αυστηρά. Αυτά τα μέτρα, ακόμα και τα πιο αποτελεσματικά, ε, δημιουργούν θέσεις απασχόλησης περισσότερες ξαναφτιάχνουμε τα σπίτια, αναδιαρθώνουμε τις επιχειρήσεις και αυτές είναι ε, επενδύσεις πάρα πολύ ε, μεγάλης έντασης εργασίας παρά τα χαζά παλιά εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας κτλ. Ε, δημιουργείται πολύ περισσότερες ε, θέσεις απασχόλησης εξοικονομώντας ενέργεια παρά ε, με τα πυρηνικά εργοστάσια. Τέλος πάντων, ε, Εμεί, ω Επιτροπή Περιβάλλοντο, μπορούμε να βοηθήσουμε την Επιτροπή βιομηχανία για αυτά τα πράγματα. Οτιδήποτε και να αποφασίσουμε για, το, για τη μείωση των εκπομπών, 20, 30, 40%, αυτό είναι σημαντικό, εξοικονόμηση ενέργεια. Και στου υπόλοιπου τύπου Ρώσοι και τα λοιπά, έφυγε βέβαια τέλο πάντων, που πιστεύουν ότι το 30% χάχα είναι απίστευτα δύσκολο και ότι δεν θα πρέπει, αποκλείεται να το, και δεν πρέπει να το βάλουμε στόχο γιατί θα μα επηρεάσει αρνητικά, δεν μπορώ να φανταστώ πώ θα οικοδομήσουμε το μέλλον μα ε, βασιζόμενοι στο φυσικό αέριο, ε, στις εισαγωγές φυσικού αερίου, στι εισαγωγέ πετρελαίου από δικτατορίε από όλο τον κόσμο. Γιατί αυτό είναι το σενάριο, αν δεν κάνουμε γρήγορα μειώσει ε, τη ε, της χρήσης των ορυκτών καυσίμων. Αυτό είναι το μέλλον. Θα είμαστε ε, εξαρτώμενοι από δικτατορε και δικτατορίε. Καλό είναι αυτό. Καλή εξωτερική πολιτική είναι αυτή. Καλή ενεργειακή πολιτική είναι. Καλή πολιτική ασφάλεια είναι αυτή. Επομένω, η συζήτηση συνδέεται και με την ασφάλειά μα. Να μειώσουμε την εξάρτηση από τα ορυκά, ορυκτά καύσιμα. Μην ξεχνάμε λοιπόν αυτή τη διάσταση. Για αυτό το δίλημα, ανάπτυξη ή μείωση των εκπομπών, θέλω να υπάρξει κάποια τροπολογία. Η μείωση των εκπομπών ε, σε συνάρτηση με την ανεργία. Αυτό το δίλημα πρέπει να μπει στην έκθεση. Η εξοικονόμηση ενέργειας επίσης και η εξωτερική πολιτική που θα αναγκαστούμε να ασκήσουμε αν δεν μειώσουμε την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα, επίσης θα πρέπει να μπει στην ε, έκθεση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούμε σε αυτό το ερώτημα. Είναι πολύ δύσκολο γιατί πρέπει να έχουμε στο νου μας τι έγινε στην Ιαπωνία και πραγματικά μιλάμε για μια καταστροφή λεχθέντων αυτών να κάνω κι εγώ κάποια σχόλια. Αν θέλουμε να πάρουμε σοβαρά αυτό το στόχο μακροπρόθεσμα, ίσως θα μπορούσαμε να μιλάμε για 20-25%. Θεωρώ ότι ο εισηγητής κάνει μια καλή πρόταση, αλλά θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι έχουμε υιοθετήσει και κατά τη διάρκεια της ημέρας έχουμε δύο εκθέσεις ε, όπου προσθέσαμε μεγαλύτερη ευελιξία στη βιομηχανία γιατί πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε σε τι συνίστανται οι στόχοι μας και ποιοι είναι οι στόχοι μας μακροπρόθεσμα. Επίσης θα πρέπει να έχουμε και μία δυνατότητα ελέγχου διαφορετικά όταν θα φτάσουμε στο μακροπρόθεσμο στόχο μα μπορεί να μας πει η βιομηχανία αυτό το τάδε ή το δίνα δεν το πράξαμε. Έτσι λοιπόν, με σοβαρό τρόπο θα πρέπει να καθορίσουμε τους στόχους και θα πρέπει να συζητήσουμε και με τη βιομηχανία. Επίσης, πρέπει να δούμε ποια θα είναι η τακτική που έχει επιλεχθεί στον τομέα των διαπραγματεύσεων. Έχουμε ήδη μια σχετική εμπειρία στην Ευρώπη και ό,τι συμβαίνει και στις άλλες ε, χώρες ε, έχει αντίκτυπο σε διεθνές επίπεδο. Θα πρέπει εδώ να δείξουμε ότι είναι δυνατό να μειώσουμε τις εκπομπές ε, και ταυτόχρονα να έχουμε και οικονομική ανάπτυξη. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα δούμε από κοινού. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη μείωση του υδραργύρου ε, μπορέσαμε να πείσουμε και τις άλλες χώρες ότι ήταν δυνατό, μπορέσαμε να κάνουμε το ίδιο και με άλλα χημικά προϊόντα, με άλλες χημικές ουσίες, ήταν δυνατό λοιπόν κάτι τέτοιο. Ακολουθούμε ένα μοντέλο σε διεθνές επίπεδο και το ίδιο πρέπει να μπορούμε να κάνουμε και σε επίπεδο κλίματος. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πώς δεν μπορούμε να πάμε πιο μακριά όταν έχουμε τόσα πρακτικά παραδείγματα θα πρέπει να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε και θα πρέπει να εργαστούμε με τον ίδιο τρόπο όταν ε, πρόκειται και για αυτά τα κλιματικά ζητήματα. Κάτι τελευταίο. Πιστεύω ότι έχουμε ένα πραγματικό πρόβλημα. Αν θέλουμε η Ευρώπη να είναι φιλόδοξη. Είναι αλήθεια ότι μπορεί να υπάρξουν προβλήματα με κάποιες βιομηχανίες ε, που ε, είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Έχουμε μιλήσει για ε, τις βιομηχανίες χάλιβα ή τις τσεμιντοβιομηχανίες. Θα πρέπει όμως να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν ισιόροι ανταγωνισμού μεταξύ αυτών των βιομηχανιών και θα μπορέσουμε να τα αναφέρουμε όλα αυτά τα θέματα και σε πλαίσιο ΠΟΕ. Σε ό,τι αφορά στα τελωνία, ξέρω ότι υπάρχουν μία σειρά προβλημάτων για πολλά κράτη-μέλη αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την προβληματική. Δεν μπορούμε να έχουμε μία κλιματική πολιτική ε, μονομερή, θα πρέπει να βρούμε λύσεις για τους διάφορους τομείς και πρέπει να είμαστε και αρκετά φιλόδοξοι. Κύριος Φλόρεντ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να πάμε προς το 30%, να πούμε δηλαδή ότι το 20% είναι δεσμευτικό και όποιος μπορεί να το ξεπεράσει και ότι τελικά ο στόχος προς τον οποίο όλοι οδεύουμε είναι το 30%. Τι κάνουμε εδώ στην Ευρώπη. Τι κάνουν τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 20-30%. Ξαφνιάζομαι γιατί βλέπω διάφοροι συνάδελφοι εδώ να μιλάνε για το 30% 40% και τα κράτη αυτά που είναι μακριά ακόμα απέχουν από το 20% δεν προτείνουν τίποτα. Εγώ κοιτάω τα νούμερα, κοιτάω τα στοιχεία, τα πραγματικά γεγονότα. Και θα προτιμούσα κύριε Πρόεδρε, αντί να μιλάμε τόσο εύκολα για αριθμούς και να λέμε 30%, να πούμε να βγει κάποιος από την πυρηνική ενέργεια. Είναι εύκολο αυτό. Το θέμα είναι πώς, πώς όμως θα πλησιάσουμε πιο πολύ στο στόχο μας που είναι αυτό το 30%. Κοιτάξτε την καταστροφή στην Ιαπωνία και βλέπετε νομίζω ότι χρειάζονται μέτρα, χρειάζονται προσπάθειες έτσι ώστε με διάφορους μηχανισμούς να φτάσουμε σε αυτό το 30% και 40% γιατί η πρόταση της Ήτρε ίσως θα πρέπει να μας οδηγήσει σε μια πιο λογική πρόταση. Δηλαδή 20 και πλέον. Και αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι πώς θα φτάσουμε προς τα εκεί. Απ' την άλλη μεριά θα ήθελα να πω ότι λυπάμαι που ο κύριος Ρώση δεν είναι πια εδώ. Γιατί δυστυχώς έφυγε, αλλά εγώ θα του εξηγούσα το θέμα των θέσεων απασχόλησης. Το θέμα αυτό αφορά καθαρά τις δομές των κρατών μελών στην ε, βόρεια Ρενανία, Βεσφαλία. Γνωρίζω καλά την περιοχή αυτή. Ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει. Σπάνε οι παλιές και απαρχαιωμένες δομές. Αυτό είτε προτείνουμε νέες τεχνολογίες είτε όχι. Ποια είναι τα κίνητρα. Ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας, αηφορία, αηφόρος ανάπτυξη. Όλα αυτά θα πρέπει να συνεχίζουμε να τα προωθούμε. Νομίζω ότι σε αυτό που μόλις ακούσαμε λείπει κάτι. Αυτό το 20% και αυτοί οι οποίοι τελικά στοχεύουν στο 30% θα πρέπει να το δούμε αν θέλετε συνολικά και ενδεχομένως να κάνουμε περισσότερες διπλωματικές προσπάθειες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε όντως να προωθήσουμε αυτό το 30%. Καταλαβαίνω. Και δεν είμαι και 100% σίγουρος ότι εγώ προσωπικά θα υποστηρίξω αυτή την πρόταση για το 30%. Αλλά δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί. Δεν μπορούμε να πούμε με ιδεολογικό και δογματικό τρόπο ότι θα πείσουμε και θα πιέσουμε όλους αυτούς που είναι στο 20 σήμερα να φτάσουν στο 30. Κύριε Ρώση, όντως είμαστε εδώ, καταλαβαίνουμε και τα οικονομικά θέματα. Είναι περίπλοκα όλα αυτά, αλλά μην ξεχνάτε ότι δύο μεγάλες, ε, δύο μεγάλοι όμιλοι, η Κρουπ και η ΔΕΣΕΦ στην ε, Γερμανία πραγματικά λειτουργούν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και βάσει των προτύπων που ε, αναφέραμε. Ναι, ναι, ναι, κύριε Φλόρενς, εγώ νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να έρθουμε σε αυτό το οικολογικό αγρόκτημα και να το επισκεφτούμε. Ναι, ναι, αυτό να το κάνουμε το καλοκαίρι στις διακοπές. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο στόχος μας είναι 20% ή 30%. Εδώ πρόκειται για μια έκθεση πρωτοβουλία. Και δεν είναι δυνατόν να βρισκόμαστε τόσο μακριά. Δεν είναι δυνατόν να πιάνουμε ή από τη μία ή από την άλλη ε, κατεύθυνση γιατί καταλαβαίνετε ότι εδώ μας έχουν οδηγήσει η Επιτροπή και το Συμβούλιο σε αυτή την κατάσταση. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλή ιδέα το 30% αν είχαμε αυτά τα εργαλεία. Το έχουμε αποφασίσει και το έχουμε ψηφίσει. Αν οι άλλοι όμως μας ακολουθήσουν. Μας ακολουθούν. Ένα μικρό βήμα έχει γίνει μέχρι τώρα. Αλλά όχι όσο σημαντικό περιμέναμε μετά την Κοπενχάγη. Είχαμε πει τότε ότι στην Κανκούν θα φτάναμε στο 50% μείωση. Είμαστε μακριά από αυτό το στόχο. Και ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε σήμερα είναι ότι η Ευρώπη θα πρέπει να παραμείνει ενωμένη και να προχωρήσει περαιτέρω. Στην Επιτροπή Βιομηχανίας είπαμε ότι οι στόχοι όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να φτάσουν τουλάχιστον το 40% και παραπάνω της 100%. Βλέπετε όμως ότι η πλειοψηφία ήταν μεγάλη. Επίσης, το θέμα της απόδοσης της ενέργειας. Πολύ συγκεκριμένος στόχος. Κύριε εισηγητά και οι σκιώδεις εισηγητές, θα πρέπει εδώ να θέσουμε στόχους από μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται, επαναλαμβάνω, για έκθεση πρωτοβουλίας. Αν δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία που ακολουθεί συγκεκριμένο lobbying. Τι θα πετύχουμε. Δεν πρέπει να παραμείνουμε μόνοι μας. Και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και στο διεθνές επίπεδο. Αυτό το 30% εμείς μπορούμε να το αποφασίσουμε εδώ. Και θα μας υποστηρίξουν όλοι, θα μας χειροκροτήσουν. Δεν θα έχουμε πετύχει όμως τίποτα. Χρειαζόμαστε μια διπλωματία ευρωπαϊκή με κεντρικό θέμα το κλίμα. Και θα πρέπει η Επιτροπή με καινούριο διαρθρωτικά διαφορετικό τρόπο να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Και βεβαίως χρειάζεται, είναι απαραίτητη η δημιουργία αυτής της υπηρεσίας της διπλωματικής, της ε, υπηρεσίας εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κεντρικό θέμα την αλλαγή του κλίματος. Και οι διεθνείς διαπραγματεύσεις μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να γίνουν. Μιλήσαμε επίσης για τους μηχανισμούς, CDM. Ήταν πολύ εξαιρετική η παρουσίαση που κάνετε στην έκθεσή σας. Και το ερώτημα μου είναι, τι αποφασίσαμε το 2008, έχει νόημα ή δεν έχει νόημα, να κάνουμε μία ανάλυση. Και αυτό βεβαίως θα μας πάρει χρόνο. Γιατί το 2008 δεν είχαμε χρόνο. Εγώ τότε την στήριξα την πρόταση. Μάλιστα πέρασε στην πρώτη ανάγνηση. Αλλά πιστεύω ότι κάποιοι συνάδελφοι που δεν είναι ούτε στη δική μας Επιτροπή εδώ, ούτε στην Επιτροπή Βιομηχανίας, υποστήριξαν χωρίς μεγάλη πεποίθηση. Και τελικά το 2009 βεβαίως εν ώψη των ευρωπαϊκών εκλογών δεν είχαμε το χρόνο που έπρεπε για να γίνει μια εις ανάλυση και συζήτηση. Αυτό πρέπει να κάνουμε σήμερα. Το 20% δεν μας αρέσει, το 30% είναι καλό και το 40% τέλειο. Ε όχι, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, δεν είναι τόσο απλή η απόφαση. Θα πρέπει καταρχήν να αποφασίσουμε για το στόχο που θέλουμε να πετύχουμε όσον αφορά τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργειας, θέλουμε να δούμε το θέμα των θέσεων απασχόληση. και θέλουμε να δούμε και τι τις διαρροές του άνθρακα. Και βεβαίως το θέμα της μεταφοράς της απασχόλησης, της μεταφοράς των θέσεων απασχόλησης από τη μία περιοχή στην άλλη και από τη μία χώρα στην άλλη. Τι μέτρα πρέπει να πάρουμε για να σταματήσει αυτό. Η στρατηγική μας για το 2020 θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να είναι στο επίκεντρο αυτής της νέας ευρωπαϊκής διπλωματικής δράσης. Η πρόθεση του Πίτερ Λίζε είναι πολύ σωστή. Δεν πρέπει να υπάρχει μια τέτοια αντιπαράθεση εδώ μέσα, σε αυτή την Επιτροπή. Αυτό το 20% ή 30% δεν μπορεί να γίνει θέμα που θα μας χωρίσει. Επαναλαμβάνω ότι αυτοί στους οποίους απευθυνόμαστε δεν πρόκειται να καταλάβουν τίποτα άλλο από το ότι είμαστε αδύναμοι σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ας στείλουμε λοιπόν ένα σαφές μήνυμα στα άλλα δύο θεσμικά όργανα, ας μιλήσουμε για το στόχο μας ε, όσον αφορά την, ε, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 40% και νομίζω ότι για τα υπόλοιπα με αυτόν τον τρόπο ενδυναμώνουμε τη θέση μας. Πρόεδρος, ωραία, θα δούμε τι θα πετύχουμε. Ναι, 20%, 30% πρέπει όμως να ορίσουμε και κάποια άλλα εργαλεία. Ο Σαλβατόρε Ταταρέλα είναι ο τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αναρωτιέμαι και ρωτώ και τους συναδέλφους. Πώς μπορούμε να φτάσουμε στα καλύτερα αποτελέσματα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Αναρωτιέμαι αν αυτό είναι δυνατό με τη συνεισφορά όλων των κρατών ή με τη συνεισφορά μεμονωμένων κρατών παγκοσμίως. και εδώ το ότι η συνδύσκευση του κακού να ήταν μια τεράστια επιτυχία. Να δούμε τις προφορικές δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις μπορώ να συμφωνήσω. Αν δούμε όμως ε, τις ε, υποχρεωτικές δεσμεύσεις που να έχουν αναλάβει τα κράτη, ούτε μία δεν βρήκα. Έτσι λοιπόν πρέπει να παραδοθούμε βεβαίω και όχι, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε που να είναι πιο σημαντικό Πιστεύω ότι το πλέον σημαντικό που μπορούμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να οθήσουμε τον υπόλοιπο κόσμο προς δεσμευτικούς στόχους. Έτσι λοιπόν στην έκθεση ένα σημαντικό τμήμα θα πρέπει να αφιερωθεί στην όθηση αυτή, δηλαδή η Ευρώπη να εργαστεί ακόμη περισσότερο από ότι στο παρελθόν για να υπάρξουν υποχρεωτικέ δεσμεύσει και από τα άλλα κράτη. Μόνο το ότι μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα αξιόλογα. Θα μετατραπούμε σε ένα διπλωματικό έθνο. Ε, όχι, αλλά πρέπει να δώσουμε και κάποιο παράδειγμα. Και όπω στο παρελθόν, δώσαμε το παράδειγμα ω Ευρώπη με αυτό το στόχο 2020. Μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτή την οδό Μπορούμε να τη βελτιώσουμε βεβαίως, ε, αλλά να είμαστε και ρεαλιστές και να λαμβάνουμε υπόψη τι συμβαίνει καθημερινά στον κόσμο. Είδαμε ότι συμβαίνουν έκτακτες ε, καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τώρα, το κύριο μειονέκτημα που βρίσκω εγώ στην έκθεση που μας προτείνεται είναι ότι φαίνεται σχεδόν να είναι ένα πολιτικό μανιφέστο. Δηλαδή ο καθένας εντάξει έχει τις ιδέες του. Αλλά φαίνεται αυτό σε ένα, ένα πολιτικό μανιφέστο που οθεί την Επιτροπή να τοποθετηθεί με ριζοσπαστικό τρόπο και να χωριστεί, ενώ ο καθένας από εμά όταν είναι εισηγητής πρέπει να προσπαθεί να βρει μία μέση οδό αποδεκτή από όλους έτσι ώστε να περάσει η έκθεση ή να μην ε, ψηφιστεί με πολύ λίγες ε, ψήφους ε, για να έχουμε θετικό πολιτικό αποτέλεσμα. Ρωτώ λοιπόν και ζητώ μάλλον από τον συγκητή να καταβάλει μια προσπάθεια να καταλάβει μια λιγότερο κάθετη θέση γιατί ξέρετε σε αυτή την επιτροπή υπάρχουν διαφορετικές ευαισθησίες ακόμη και στο εσωτερικό των ομάδων. Πρέπει λοιπόν ε, να υπάρχει ένα πνεύμα ανοιχτό στο συμβιβασμό προκειμένου να μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τις θέσεις των άλλων. Δηλαδή δεν αναφέρεται καθόλου η έκθεση στον οδικό χάρτη της Επιτροπής. Θα έπρεπε να αναφέρεται αυτό. Δεν αναφέρει η έκθεση μέσα σαφήνεια τα μέσα τα εργαλεία με τα οποία αυτά τα επιθυμητά φυσικά αποτελέσματα θα μπορούσαν να επιτευχθούν. Η έκθεση δεν ε, θέτει το πρόβλημα του οικονομικού αντίκτυπου. Ε, αντίθετα, παρουσιάζει ένα, παρα, ένα ε, σενάριο που αντιστοιχεί σε ένα παράδεισο, ότι δηλαδή θα βελτιώσουμε την υγεία, τι θέσει εργασίας κτλ. Όμως εγώ νομίζω ότι υπάρχουν ε, και κάποιε συνέπειες και μία ανάλυση εις βάθος επί των συνεπειών ε, θα ήταν κάτι που θα μπορούσαμε να δεκτούμε. Υποβάλλω λοιπόν εδώ αυτές τις προτάσεις στον συγητή. Όλοι θα υποβάλουμε τροπολογίες, αλλά τελικά πρέπει να καταλήξουμε σε έναν αποδεκτό συμβιβασμό. Σε αυτή την επιτροπή πολύ συχνά υπογραμμίζεται με ιδιαίτερη έμφαση ο στόχος να έχουμε ένα καλύτερο κλίμα για ένα καλύτερο περιβάλλον. Βεβαίως έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι στον κόσμο προκύπτουν και έκτακτες καταστάσεις και ε, θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις με πιο φιλόδοξο τρόπο. Μιλώ για την καταστροφή που έλαβε χώρα στην εμπονία αυτές τις μέρες. Μιλώ για την πείνα, για την ανέχεια, για την ειρήνη, για την απασχόληση. Έχουμε δραματικά γεγονότα και θα έπρεπε να προσδώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ακούσαμε πολλά επιχειρήματα. Θα ακούσουμε την Επιτροπή. Και κατόπιν ε, θα πάρει το λόγο ο εισηγητής. Ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή και όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πολύ καλή έκθεση και την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχω κάποιε παρατηρήσει και θα προσπαθήσω να απαντήσω και σε ορισμένα ερωτηματικά που τέθηκαν. Το πρώτο σχόλιο μου είναι αυτό με το οποίο ξεκίνησατε και εσείς Πρόεδρε, ότι η κλιματική αλλαγή και η δράση για το κλίμα δεν ε, είναι θέματα που αφορούν μόνο το περιβάλλον, αλλά και οικονομικά και βιομηχανικά ζητήματα και συνδέονται ιδιαίτερα με το πώς ε, βλέπουμε την ε, μελλοντική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Γι' αυτό ε, σε πολύ καλή χρονική στιγμή έρχεται αυτή η συζήτηση. Η Κομισιόν την περασμένη εβδομάδα δημοσίευσε τον οδικό χάρτη μέχρι το 2050 και το πιο σημαντικό μήνυμα που ήρθε από τον οδικό χάρτη είναι η σαφή επιλογή που έχουμε ω εξή, αν ακολουθήσουμε την οδό τη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, σημαίνει ότι θα επενδύσουμε στην εγχωρή οικονομία και προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε και αριθμητικά στοιχεία. Φυσικά είναι βέβαια τα οικονομικά στοιχεία γιατί έχουμε μακροπρόθεσμη προοπτική. Όμω, ε, πρέπει να δούμε ότι πρέπει να γίνουν πολύ μεγάλε επενδύσει σε διάφορου τομεί ηλεκτρική ενέργεια, αυτοκινητοβιομηχανία κτλ. στην εγχώρια οικονομία μα, αλλά θα έχουμε και εξοικονόμηση στα καύσιμα αν ε, προβούμε σε αυτές τις επενδύσεις. Αυτό είναι το σημαντικό μήνυμα από τον οδικό χάρτη. Και ένα δεύτερο μήνυμα από τον οδικό χάρτη σχετικό για τη συζήτηση αυτή είναι το εξή. Εξετάσαμε διάφορα σενάρια για το πόσο γρήγορα πρέπει να πάμε για να πετύχουμε τους στόχους του 2015 και το μήνυμα που έχουμε εκεί είναι ότι το 25% της εγχώριας μείωσης ε, είναι ε, μία οδός που μπορεί να μας οδηγήσει στο 80% μείωση για το 2050 με αποτελεσματικό τρόπο προς το κόστος. Η οικονομική ανάλυση μας έδειξε ότι αν κάνουμε λιγότερα τα επόμενα 20 έτη, τότε θα μας κοστίσει περισσότερο αργότερα. Δεύτερο σχόλιο. Πολλοί βουλευτέ τοποθετήθηκαν για το θέμα των διεθνών διαπραγματεύσεων και ότι πρέπει να σημειώσουμε μεγαλύτερη πρόοδο. Όλοι συμφωνούμε από αυτό και εργαζόμαστε σκληρά στι διεθνεί διαπραγματεύσει. Θέλω να τονίσω ότι η σημερινή κατάσταση διαφέρει πριν ε, τρία έτη όταν ε, υιοθετήσαμε τη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια. Ήταν μονομερή σε στόχο, και η Κομισιόν ήθελε να δείξει ηγετική θέση ενάντια τη Κομεχάγη, πρώτη Κομεχάγη σήμερα οι ηγέτε στο Κανκούν και στην Κοπενχάγη έχουν ε, υιοθετήσει το στόχο των δύο βαθμών και επίσης υπάρχει και δέσμευση από πάνω από 80 χώρες και μάλιστα από μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες στον κόσμο να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση. Και αυτό διαφέρει από το πρωτόκολλο του Κιώτο, το οποίο έθετε δεσμευτικούς στόχους για τις αναπτυγμένες χώρες. Τώρα βλέπουμε την Ινδία, την Κίνα, την Βραζιλία, την Νότια Αφρική να αναπτύσσουν συγκεκριμένα σχέδια και να εφαρμόζουν ε, τις δεσμεύσεις, τις υποσχέσεις που έχουν κάνει. Ε, πρόσφατα και το πενταετές έτος σχέδιο, μας συγχωρείτε, της Κίνας και όποτε φαίνεται η Κίνα θέλει να σεβαστεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και καταβάλει προσπάθειες για να αναπτύξει νέες τεχνολογίες μέσω της καινοτομίας σε πολλούς τομείς. Το θέμα για τη διπλωματία. Η κυρία Άστον έχει αναλάβει αυτή τη δέσμευση, αλλά φυσικά και η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, θα έχει τέτοια καθήκοντα. Έτσι λοιπόν θα ενισχύσουμε τις προσπαθίες μας ε, για να προωθήσουμε τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για τη διαρροή του άνθρακα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας Πιστεύω το σημαντικό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι στη δέσμη μέτρων για το κλίμα και για την ενέργεια ήταν ένα από, τα, από τους κύριους πυλώνες και ε, το συμβιβασμούς μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου που σήμερα εφαρμόζουμε πολύ συγκεκριμένα με benchmarking και αναδιανομή και θέλουμε να αποφύγουμε τη μελλοντική διαρροή άνθρακα. Έχουμε λοιπόν την ελεύθερη διανομή και έχουμε τη δυνατότητα να καταπολεμήσουμε έμεσα την έμεση διαρροή του άνθρακα. Τώρα, αυτό που εξετάσαμε εκ νέου στον ε, οδικό χάρτη και στην οικονομική ανάλυση για το 2050 είναι αν επαρκούν όλα αυτά τα μέτρα. Βασικά λέμε ότι έχουμε δύο αντικειμενικού λόγους για του οποίου είναι χαμηλότερη κίνδυνη από ότι στο παρελθόν όταν ευθύσαμε το πακέτο για την ενέργεια και το κλίμα. Ένα, είναι χαμηλότερε οι τιμέ του άνθρακα. Δεύτερον, Άλλες χώρες όντως εφαρμόζουν και έχουν θετήσει τις δεσμεύσεις της Κοπενχάγης, τις υποσχέσεις της Κοπενχάγης. Έτσι λοιπόν υπάρχουν δεσμεύσεις και από την άλλη πλευρά για δύο συγκεκριμένα τώρα ζητήματα. Υπήρχε μια ερώτηση για τη σχέση με την ατμοσφαιρική ρήπανση. Κύριος Ρώση. Ε, η δράση για την κλιματική αλλαγή σημαίνει η μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα και χρησιμοποίηση ε, καθαρότερων εναλλακτικών τεχνολογιών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχουν αντίκτυπο ε, στους ρηπογόνες ουσίες, ε, στους ρήπους που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα. Έτσι λοιπόν αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα καθαρό όφελος και προσπαθούμε αυτό να το προσωπικοποιήσουμε στην ανακοίνωσή μας. Τέλος, είχαμε και μια ερώτηση από τον κύριο Ντέιβις ε, για ε, ποιος θα ήταν ο αντίκτυπος ε, στις τιμές του άνθρακα. Πρέπει να το εξετάσει η Κομισιόν αυτό περαιτέρω, αν εξετάσει το θέμα του SETA site. Στον οδικό χάρτη εξετάσαμε τις σχέσεις μεταξύ του σχεδίου εκπορίας εκπομπών και των ενεργειακών πολιτικών. Είτε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ETS, το σχέδιο εκπορίας εκπομπών και το set site για να δώσουμε καλύτερα κίνητρα για ενεργειακή αποδοτικότητα, γιατί το ίδιο το SETA site ε, θα έδινε ισχυρότερα κίνητρα στις εταιρείε και στις βιομηχανίες ε, να βελτιώσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα. Έτσι λοιπόν αυτό θα είχε αποτέλεσμα και στην κυρία Νικίνωση λέμε ότι προκειμένου να φτάσουμε στο 30% δεν το λέμε αυτό στο οδικό χάρτη αλλά στην περίπτωση που θα πάμε στο 30% θα πρέπει να ε, δέσουμε κατά μέρος δικαιώματα 1,4 δις δηλαδή από 30 θα πάμε στα 60 ευρώ αλλά αυτό το, ε, το set aside σημαίνει ότι θα αξιολογήσουμε ποια μέτρα θα πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή στον τομέα της ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ για τις εξηγήσεις σας. Ο εισηγητής τώρα. Uh, Ευχαριστώ. Θα είμαι ξεκάθαρος από την αρχή. Δεν θέλω να με χειροκροτήσετε ε, για την υλοποίηση ενός στόχου. Και κύριε Ταταρέλα, δεν θέλω να διχάσω το κοινοβούλιο. Ε, αυτή η συζήτηση κρατάει εδώ και καιρό. Συνεχίζεται και συμφωνώ με κάποιους από τους συναδέλφους που είπαν ότι είναι μια θεμελιώδη συζήτηση για την κατεύθυνση που θα πρέπει να κάνει η οικονομία. Αυτή η συζήτηση θα πρέπει να γίνει. Τελικά θα ληφθεί μια πολιτική απόφαση για ένα ποσοστό. Εγώ δεν θέλω όμως χειροκροτήματα. Καθώς θέτω το ποσοστό, δεν επιζητώ τα ε, χειροκροτήματα. Το θέμα είναι να γίνει αυτή η συζήτηση και στο τέλος θα γίνει και μια, θα ληφθεί και μια απόφαση, ένα πολιτικό συμπέρασμα για το ποσοστό. Ε, επίσης, δεν είναι πολιτικό μανιφέστο των Πρασίνων, ε, γιατί αν θέλετε να διαβάσετε πραγματικό πολιτικό μανιφέστο των Πρασίνων, ε, είναι πολύ πιο δεσμευτικό και στεναρό. Ε, όσοι με ξέρουν και έχουν ε, συνεργαστεί μαζί μου, ξέρουν ότι μου αρέσουν οι συμβιβασμοί. Θέλω να μιλήσω για το διεθνέ πλαίσιο, για τι μετεκαταστάσει των επιχειρήσεων και για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Για το διεθνέ πλαίσιο. Συμφωνώ ότι κάτι θα πρέπει να πούμε για αυτό το θέμα. Να μιλήσουμε για την κλιματική διπλωματία, γιατί για το κλίμα είναι σημαντικό όλο ο κόσμο να κάνει κάτι και όχι μόνο η Ευρώπη. Όμω, αυτή τη φορά η συζήτηση αλλάζει ρότα. Αυτή τη φορά θέλω να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό που κάνουμε θέτοντας αυτού του στόχους στην Ευρώπη είναι κάτι παραπάνω από τη βιομηχανική πολιτική. Δεν εξαρτώμαστε πια από τις διεθνείς διαπραγματεύσεις, είναι το τι θέλουμε να πετύχουμε εμείς στην Ευρώπη. Τι είδους οικονομία θέλουμε να φτιάξουμε. Και επομένως, ναι, για τους κλιματικούς στόχους, ο υπόλοιπος στόχος πρέπει να κουνηθεί. Αλλά πέρα από αυτή τη συζήτηση είναι σημαντικό να δούμε τι θα πετύχουμε εμείς ως Ευρώπη μόνοι μας. Η Κίνα είπε πολλές φορές, φορές το εξή. Να σα το πω ξεκάθαρα. Αν υπάρχει μία χώρα η οποία θα υποφεληθεί από τις καθυστερήσεις της διεθνής διαπραγματεύσεις θα είναι η Κίνα. Η Κίνα έχει μια ταχαίως αναπτυσσόμενη οικονομία, ε, έναν πληθυσμό που αυξάνεται, ε, το εκπαιδευτικό σύστημα πλαταίνει και αυξάνεται. Θέλουν λοιπόν να βυθίσουν όλες τις διεθνείς διαπραγματεύσεις, γιατί ξέρουν ότι αυτές οι καθυστερήσεις τους βοηθούν. Είναι υποφελής για αυτούς και όχι για την Ευρώπη. Εμείς είμαστε στην πρωτοκαθεδρία της τεχνολογίας. Αν θέλουμε να κρατήσουμε αυτή τη θέση όμως πρέπει να κουνηθούμε, γιατί πέρυσι ήταν ξεκάθαρο ότι η Κίνα είναι το νούμερο ένα για, στο δίκτυ α, βιώσιμων επενδύσεων. Οι Ernest Young κάνουν αυτές τις α, βαθμονομήσεις και η Κίνα είναι πρώτη. Επομένως κουνιέται η Κίνα. Εμείς χάνουμε ως ε, Ευρώπη και αν δεν κάνουμε τίποτα θα χάσουμε κι άλλο. Επομένως, ναι, η κλιματική διπλωματία σημαντική, αλλά μην ξεχνάτε τι θέλουμε να πετύχουμε ως Ευρώπη. Τώρα, το ενδεχόμενο μετεγκαταστάσεων. Κύριε Ρώση, ε, δεν πιστεύω ότι η γη είναι επίπεδη. Έτσι, κύριε Ρώση. Καλό να σας το πω να τα ακούσετε. Και, ναι, είμαι ανοιχτό στου συμβιβασμού. Αλλά όμως να κάνουμε συμβιβασμού μετά από επιχειρήματα. Γιατί ξέραμε ότι την πρώτη περίοδο ε, υπήρχαν μεγάλα κέρδη για την ε, βιομηχανία. Ε, κερδίσανε χρήματα από το ETS, από το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι έχουν και για την τρίτη περίοδο, ας πούμε, δωρεάν εκπομπές. Ε, υπάρχουν και διαρροές του άνθρακα. Δηλαδή, αυτές οι δωρεάν εκπομπέ δεν τους κοστίζουν τίποτα. Και τρίτον, φέτος θα επιβάλλουμε ε, κρατικές κατευθυντήριες γραμμές, όπου κρατικές ενισχύσεις μάλλον, κατευθυντήριες γραμμές για τι κρατικέ ενισχύσει. Ασχολούμε με αυτό το θέμα του, της διαρροής του κεφαλαίου σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο Σημαντικό είναι και αυτό, αλλά μην ξεχνάμε και το περιεχόμενο. Ξέραμε μέχρι στιγμή ότι οι κλιματικέ πολιτικέ δεν οδήγησαν σε μεγάλε δαπάνε στην ε, βιομηχανία, αντίθετα κέρδισαν από αυτήν την ιστορία. Εάν θέλουμε λοιπόν να μιλήσουμε για γεγονότα, να μιλήσουμε. Έτσι. Και να μιλήσουμε για ένα κόσμο που δεν είναι επίπεδο, για μια γη που δεν είναι επίπεδη. Λοιπόν, ενεργειακή αποδοτικότητα. Τελευταίο κεφάλαιο, ε, τον έφεραν διάφοροι. Προφανώ θέλω να συμβιβαστούν να συμβιβαστούμε με τροπολογίες, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα, γιατί ναι, είναι τεράστια σημασία. Και όπως είπε και η Κομισιόν σήμερα, εάν πετύχουμε τους στόχους της ενεργειακής αποδοτικότητας, τότε ήδη έχεις πετύχει εγχωρίως ένα στόχο του 25%. Το επαναλαμβάνω, εγχώριο στόχος. Αυτό το είπε η Κομισιόν, το είπε σήμερα, ακόμα μια φορά. Τώρα, αν θέλουμε να πετύχουμε πραγματική ενεργειακή αποδοτικότητα, θα πρέπει να προσαρμόσουμε ε, τους στόχους μας στα πλαίσια του συστήματος εμπορίας απομπών και εκτός. Γιατί αν μια χώρα επενδύει στην ενεργειακή αποδοτικότητα, μια χώρα άλλη, αν δεν προσαρμοστούμε, να αγοράσει. Επομένως, θα πρέπει να προσαρμόσουμε τους στόχους, ούτω ώστε να αδράξουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα. Αλλιώ λέμε, εντάξει, εθελοντικέ συμφωνίε, μπορούμε να σπρώξουμε για ενεργειακή αποδοτικότητα, αλλά επί της, ουσία, επί της ουσίας δεν θα έχουμε λιγότερες εκπομπές, απλώς προσαρμόζουμε τους στόχους. Γι' αυτό πρέπει να ευθυγραμμίσουμε το σύστημα εμπορίας εκπομπών, το ETS και, τα, και το τι συμβαίνει εκτός ETS. Καταληκτικά, ναι, θέλω, φίλοι μου, να συμβαστώ σε τροπολογίε, δεν θέλω να διχάσω το κοινοβούλιο, θέλω να γίνει η συζήτηση με πραγματικά επιχειρήματα, με επιστημονικά επιχειρήματα και μετά να περάσουμε στις πολιτικές δηλώσεις. Είναι μια ουσιαστική συζήτηση. Πρέπει να δούμε πού πιστεύουμε εμείς ότι πρέπει να κινηθεί η ευρωπαϊκή οικονομία. Θα υπάρξει τελικά πολιτικός, πολιτική απόφαση για το στόχο. Ε, ξέρω ότι θα υπάρξουν άλλοι στόχοι για το 2050, αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε στο 2020. Ε, και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν μπορούμε να ξεχάσουμε αυτή τη συζήτηση, δεν μπορούμε να τη βάλουμε στο περιθώριο. Ευχαριστώ και περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία και με ανοιχτό πνεύμα τη συζήτηση. Και ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχω ένα, μια σημαντική ανακοίνωση να σας κάνω. Καταρχάς, η Λίντα Μακάβεν, ένα διαδικαστικό. Δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέλω να πω. Μιλάμε για την ε, εξοικονόμηση ενέργειας. Ε, το δωμάτιο όλο και ψυχραίνει. Έχω ψοφίσει στο κρύο. Ε, εντάξει, να μην να μην ε, δαπανάμε ας πούμε, ενέργεια με το καλοριφέρ, αλλά μην βάζουμε και κλιματισμό το Μάρτιο, έτσι. Ε, έχω την αίσθηση ότι εδώ πέρα έχουμε τον κλιματισμό με κρύο αέρα. Ελπίζω οι τεχνικοί μας να μας ακούνε. Λοιπόν, παίρναμε στη σημαντική ανακοίνωση όπως σας προανήγγυλα. Η κατάθεση των τροπολογιών είναι μέχρι τις 24 Μαρτίου στις 12 και όχι στις 25 Μαρτίου, όπως λέει το κείμενό σας, έτσι. Τελική ημερομηνία 24 Μαρτίου μεσημέρι, 12 η ώρα. Η γραμματεία θα σας στείλει και ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ούτως ώστε οι βουλευτέ, οι οποίες είναι απόντες να μάθουν ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι 24η Μαρτίου. Και τώρα θα πάμε στο επόμενο σημείο, είναι η τροποποίηση του κανονισμού 1406 του 2002 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Ο εισηγητή μα είναι ο κύριο Στάση. Του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Πολύ θα θυμάστε την, καταστροφή του Έρικα και την ε, πετρελοκυλίδα που προέκυψε. Επίσης, έχουμε ένα σχέδιο κανονισμού τώρα. Έχουμε ένα κανονισμό, είχαμε μάλλον ένα κανονισμό, ο οποίος τροποποιείται τώρα ε, αυτός ο κανονισμός ε, δημιουργήθηκε λόγω αυτής της πετρελοκυλίδας και μάλιστα γι' αυτό δημιουργήσαμε και την, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Θάλασσας, ο οποίος λειτουργεί το 2003. Έκτοτε ο κανονισμός τροποποιήθηκε τρεις φορές. Ε, μετά την κρίση επίσης ε, του Πρεστή, το 2002 εξασφαλίσαμε ότι ο οργανισμός αυτός ο ΕΜΣΑ θα έχει μια σειρά από νέα καθήκοντα μεταξύ άλλων θα έχει την αρμοδιότητα για αυτές τις καταστροφές. Η ΕΜΣΕ επίσης επιθεωρεί και τα πετρελαιοφόρα σκάφη. Θα θυμάστε την πλατφόρμα εξόριξης πετρελαίου στον κόλπο του Μεξικού και την καταστροφή επίσης στον κόλπο του Μεξικού. Η Κομισιόν αντέτρασε γρήγορα. Ο Επίτροπος Έτιγκερ εμφανίστηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και μίλησε μετά από το ατύχημα. Κάναμε συζητήσει στην Ολομέλεια, αναγκάσαμε την Κομισιόν να συντάξει μία ανακοίνωση και υιοθετήσαμε ομόφωνα ένα ψήφισμα στο Κοινοβούλιο ε, όπου αναλύαμε όλα όσα πρέπει να γίνουν για αυτές τις υπεράκτιες εξέδρες εξόρυξης πετρελαίου και τις εγκαταστάσεις τους. Και ένα από τα συμπεράσματα στο οποίο φτάσαμε είναι ότι ο κανονισμός του Οργανισμού ε, Προστασίας της Θάλασσας θα πρέπει να τροποποιηθεί. Γνωμοδοτούμε ε, στην, ε, στην έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών. Ε, λόγω της σημασίας που έχει η όλη συζήτηση για την καταστροφή του κόλπου του Μεξικού. Η δουλειά μου εδώ είναι να εξασφαλίσουμε ότι τις συστάσεις μας θα τις μετατρέψουμε σε, σε συμπεράσματα και ότι θα προκύψουν αλλαγές στην νομοθεσία από αυτές. Έχουμε 8 τροπολογίες ε, στο διατακτικό, 6 στα εκτιμώντας και 14 όπου μεταξύ αυτών υπάρχει μία ομάδα τροπολογιών που αφορούν την επέκταση του πεδίου του καονισμού ΕΜΣΑ για να, κατα... για να καλύψει και αυτές τις περάκτιες εξέδρες. Ε, δύο τροπολογίες που είναι φυσικό αποτέλεσμα της επέκτασης ε, του, της εμβέλειας. Αν συμπεριλάβουμε και τις υπεράκτιες εξέδρες, τότε οι ευθύνες του διευθυντή θα πρέπει να αλλάξουν Επίσης, αν επεκτείνει το έργο του Οργανισμού Αυτοπροστασίας της Θάλασσας, του ΕΜΣΑ, και αυτό το έβαλε σε εκτιμώντα όχι σε άρθρο, τότε πρέπει να δούμε και τις συνέπειες για τον προϋπολογισμό και το προσωπικό. Επίσης, ε, επιτρέπουμε τις επιθεωρήσεις σε τρίτες χώρες και στην Μεσόγειο και στην Μαύρη Θάλασσα, γιατί και εκεί υπάρχουν τέτοιες εξέδρες ε, υπεράκτιες. Το 11, ας πούμε, μιλάει για τη, ο, η τροπολογία 11 μιλάει για τη χρήση του δορυφορικού συστήματος που είναι στη διάθεση της ΕΜΣΑ για να δει αν υπάρχουν διαρροές πετρελαίου και αν τις εντοπίσει. Να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν το δορυφορικό σύστημα για να δούμε ε, ενδεχόμενες διαρροές από αυτές τις υπεράκτες ε, ε, εξέδρες. Ε, υπάρχει μια άλλη ομάδα τροπολογιών, μια δημόσια ερώτηση ουσιαστικά είναι αν κάνει επιθεωρήσεις, ή μάλλον κάνει επιθεωρήσεις η Κομισιόν και υπάρχουν κάποιες εκθέσεις που προκύπτουν από αυτές τις εκθέσεις και θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν και ηλεκτρονικός πώς. Άλλη ομάδα, δύο, αφορά την πολιτική αδειών γιατί η ΕΜΣΑ έχει δικοδομήσει μια εμπειρία. Η Κομισιόν θα πρέπει να υποβοηθηθεί ε, από την ΕΜΣΑ για την εκχώρηση των αδειών, για να εντοπίσει την παραγωγή πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Άλλη ομάδα ε, τροπολογιών, δύο ουσιαστικά, αφορά το σύστημα ε, ταυτοποίησης της, του οργανισμού. Αυτό θα πρέπει να αφορά όχι μόνο τα σκάφη μεταφέρουν πετρέλαιο, αλλά και άλλα σκάφη. Αυτό θα μπορούσε ε, να αξιοποιήσει και την τεχνική που έχει στη διάθεσή της ο οργανισμός. Υπάρχουν ε, και κάποιοι σκιώδεις εισηγητές που με υποστηρίζουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Ε, ελπίζω να με υποστηρίξουν και βουλευτές, οι οποίοι βέβαια δεν υπάρχουν, διότι η αίθουσα είναι κενή. θέλουν να πάνε να φάνε. Ε, Ευχαριστώ, Μπάρτ. Έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μα. Έτσι λοιπόν θέλω να ζητήσω από όλου του σκιώδει εισηγητέ να προσπαθήσουν να περιοριστούν στα δύο λεπτά. Κυρίω ε, ο σκιώδη εισηγητή του ΕΛΚ. Η σκιώδη εισηγητρία του ΕΛΚ, μάλλον. Νομίζω ότι οι σκέψεις του εισηγητή είναι καλές, είναι λογικές και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί άκουσα ότι οι νομικές πράξεις που ρυθμίζουν τη δράση της ΕΨΑ έχουν ολοκληρωθεί. Στηρίζω λοιπόν την, τον ε, εισηγητή της γνωμοδότησης Ιδιαίτερα όταν λέει ότι πρέπει να καλυφθούν και οι πλατφόρμες offshore, εξόρυξης πετρελαίου, ότι πρέπει δηλαδή να καλύπτονται και αυτές. Αυτό που είναι σημαντικό βεβαίως τώρα να δούμε είναι τι προβλέψεις υπάρχουν και αν καλύπτονται και οι μεταφορές. Γιατί ξέρω παραδείγματος χάρη ότι σε περιπτώσεις όπου το φυσικό αέριο ε, μεταφέρεται κάτω από τη θάλασσα με αγωγούς. Δεν νομίζω να καλύπτεται και αυτή η περίπτωση. Εδώ βεβαίως ξέρω ότι έχει υπάρξει συνεργασία με την Νορβηγία και την Ισλανδία. Ίσως θα πρέπει να βρούμε και άλλες χώρες. Υπάρχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες αυτού του οργανισμού και θα πρέπει ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός κρατών να συνεργαστεί. Υπάρχει η Μεσόγειος, υπάρχει η Μαύρη Θάλασσα, αλλά δεν πρέπει να περιοριστούμε μόνο σε αυτή, πρέπει να πάμε και στις Βόρειες Θάλασσες και στην Όστσε. Γιατί και εκεί υπάρχουν πολλές πλατφόρμες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή έκθεση, μια πολύ καλή γνωμοδότηση και σε μεγάλο βαθμό στηρίζω αυτές τις προτάσεις και για τον οργανισμό αλλά και για το πώς στο μέλλον μπορούμε να επεκτείνουμε τις αρμοδιότητες ε, του οργανισμού αυτού. Έχω μία ερώτηση. Κάτι που βεβαίως απασχολεί ιδιαίτερα και την Επιτροπή Μεταφερών μπορεί να φτάσουμε κάποια μέρα σε μια ευρωπαϊκή ακτοφυλακή. Αυτό το θέμα το έχουμε ξανασυζητήσει στο Κοινοβούλιο, αλλά προκύπτει και στα πλαίσια αυτής της έκθεσης. Και ξέρω ότι βεβαίως οι αρμοδιότητες ε, της, ε, του φορέα αυτού, του οργανισμού αυτού, θα πρέπει ενδεχομένως να επεκταθούν και προς αυτή την κατεύθυνση. Η Επιτροπή Μεταφορών σίγουρα ε, ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό. Αν πραγματικά θέλουμε να ελέγξουμε, αν θέλουμε να υπάρξουν έλεγξη, τότε πραγματικά θα πρέπει να δούμε τι αρμοδιότητες χρειάζονται. Είναι βεβαίως μετά προκύπτουν θέματα χωρικών υδάτων, ε, συνόρων, ε, πράγματα που στο δίκαιο ε, των θαλασσών θα πρέπει να καθοριστούν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά πιστεύω ότι η αρμοδιότητα της ΕΜΖΑ θα πρέπει εδώ να επεκταθεί. Ευχαριστώ. Θέλω να πάω στον συγκεκριτή ότι εκτιμώ την εκθεσή του. Δεν έχω ειλικρινά πολλά να προσθέσω, θα είμαι γρήγορη λοιπόν. Θα είμαι σύντομη. Για το πρόβλημα για τις πλατφόρμες δεν έχει εξαφανιστεί, για τις υπεράκτες εγκαταστάσεις. Αναμένω την έκθεση της Επιτροπής για το θέμα αυτό. Ακόμη δεν έχουμε λάβει το σχετικό έγγραφο όσο το συντομότερο το λάβουμε, τόσο το καλύτερο. Δεύτερον, ε, υπογραμμίζω την επέκταση της ε, των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού έτσι ώστε να καλύπτονται και περάκτες εγκαταστάσεις εξόρξης και παραγωγής αερίου και πετρελαίου. Ε, το ψηφίσαμε τον Οκτώβριο του 2010, έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες του οργανισμού και πρέπει τα μέσα της να αυξηθούν για ε, και πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί να μην δίνουμε αρμοδιότητες σε οργανισμούς που δεν μπορούν να τις ε, ασκήσουν. Επίσης, ε, πρέπει ο οργανισμός να βοηθήσει την Κομισιόν για την, για παρακολούθηση των περιοχών στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο, αλλά και σε περιοχές όπου έχουμε εξόριξη και πιστεύω ότι η προγνωμοσύνη του οργανισμού για την καταπολέμηση των ατυχημάτων στη θάλασσα μπορεί να είναι κάτι πολύ χρήσιμο ε, μέσω και παρακολούθησης των συμφωνιών για την εξόριξη και την παραγωγή πετρελαίου και αερίου. Πρόεδρος. Δεν βλέπω εδώ ούτε τον κύριο Φερέα, ούτε τον κύριο Στίβενς. Έτσι λοιπόν, κανένας άλλος και ο δεν είναι εδώ. Ολοκληρώνεται λοιπόν συζήτηση. Αλλά νομίζω ότι ο κύριο Οικονόμου θέλει να πάρει το λόγο ξανά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τι προτάσει που σας παρουσίασα και για την εισαγωγή του. Θα ήθελα να σχολιάσω κάποιες από τις ε, τροπολογίες από την πλευρά της Κομισιόν. Φυσικά κατανοούμε το πόσο ευαίσθητο είναι το θέμα των εγκαταστάσεων εξόρυξης ε, πετρελαίου και αερίου και γι' αυτό στην πρότασή μας έχουμε εισαγάγει τη δυνατότητα να παρέμβει ο ΕΜΣΑ για να αντιμετωπίσει την ρήπανση που προκαλείται από αυτές τις πηγές. Παρ' όλα αυτά, αυτό που ζητάτε τώρα με μια σειρά τροπολογιών του εισηγητή είναι να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Και ο ΕΜΣΑ να εποπτεύει, να επιθεωρεί ε, αυτές τις πλατφόρμες προκειμένου να προλαμβάνει τη ρήπανση. Όπως γνωρίζετε, ετοιμάζουν οι υπηρεσίες Κομισιόν Ανάληψη Δράσης ε, σε αυτό το τομέα. Έτσι λοιπόν είναι κάπως αδέξιο να ζητάτε από ένα κοινοτικό οργανισμό να παρέμβει πριν να έχουμε συστήσει έτσι λοιπόν, να σας υπενθυμίσω ότι οι θεωρήσεις ε, που υλοποιεί ο ΕΜΣΑ σε άλλους τομείς που διευκρινίζονται στον κανονισμό, βασίζονται σε νομικές βάσεις, όταν ε, έχουμε παραδείγματο χάρη την επιθεώρηση κάποιων οργανισμών εταιριών ή άλλων οργανισμών σε τρίτες χώρες. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ πλοκό το θέμα πώς θα μπορούσε ο να παρέμβει σε τρίτες χώρες ε, κάνοντας επιθεωρήσεις. Αυτή την ανησυχία ήθελα να εκφράσω από τη δική μου πλευρά. Επίσης, να διευκρινίσω ορισμένα σημεία σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες 4 και 10. Γιατί ο εισηγητής αναφέρει εκεί ότι τα σημερινά συστήματα εποπτείας μέσω της ΕΜΣΑ αφορούν ε, μόνο τα δεξαμενόπλια ε, τα πετρελαιοφόρα. όμως θέλω να σας πω ότι αφορούν όλα τα πλοία που είναι άνω μια συγκεκριμένη χωρητικότητα. Αυτό λοιπόν ήδη καλύπτεται. Και ε, ίσως αν χρειαστεί να σας δώσω και περαιτέρω εξηγήσεις διμερώς. Επίσης, να αναφερθώ και στην πρότασή του για περαιτέρω διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις επιθεωρήσεις που δεν γίνονται από την ΕΜΣΑ. Να δηλώσω ότι η Κομισιόν ε, θεωρεί ε, ότι τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων ε, τροφοδοτούν τη θεσμική δουλειά της Κομισιόν για την προετοιμασία ανάληψης δράσης στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα λοιπόν και βοηθά την Κομισιόν στο να ελοπίσει το δικό της έργο. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Συγητής έχει το λόγο για τελικά σχόλια. Ευχαριστώ. Εδώ βλέπουμε ότι ε, ίσως να υπάρχει ένα μικρό νομικό πρόβλημα εδώ ή εκεί, όμως πρέπει να το συζητήσουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή, το έχουμε σκεφτεί και θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε μια τέτοια συζήτηση. Όμω, καταρχήν θα ήθελα να γίνει μια συζήτηση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφαλεία στη Θάλασσα. Είμαι έτοιμο να κάνω αυτό το βήμα παρουσιάζοντας τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση για την Ευρωπαϊκή Εκτοφυλακή και να συζητήσουμε και με την Κομισιόν για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρουσα συνεισφορά από τη δική μας πλευρά. Ευχαριστώ πολύ. Προθεσμοί για τις ε, τροπολογίες 24 ε, Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι. Η ψηφορία προβλέπεται προβλέπεται 19 Απριλίου. Καλή σας όρεξη και θα τα ξαναπούμε στις 3 ακριβώς.